Good afternoon. Καλησπέρα. Κυρίες και κύριοι μου, αγαπητοί δε συνάδελφοι, συνάδελφοι, παρακαλώ καθίστε, γιατί σε λίγο θα αρχίσουμε. Είναι η απογευματινή συνεδρίαση της Επιτροπής ΕΛΕΦ και προβλέπει ψηφοφορίες. Παρακαλώ λοιπόν να προσέχετε την κάρτα σας. Την ηλεκτρονική σας κάρτα εννοώ. Όλοι έτοιμοι. Στο... Φύγαμε. We have three votes to go. Έχουμε τρεις ψηφοφορίες. Τρεις. Η δεύτερη θα είναι και η δυσκολότερη. Ας αρχίσουμε όμως από την πρώτη. Δηλαδή η έγκριση των συστάσεων των συντονιστών. 24 Απριλίου συνεδρίασαν και μάθαμε ότι υπήρχε μια πρόταση για την Ολομέλεια στην Σύνοδο του Μαΐου για τη συμπερίληψη συζήτησης για παράνομες πρακτικές στην Βουλιγαρία. Επιτήρηση δηλαδή πολιτικών και δημοσιογράφων. Η διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε να μην συμπεριληφθεί αυτή η συζήτηση στην Ολομέλεια, αλλά το θέμα να παραπευθεί στην Επιτροπή ΕΛΕΦ. Και την ίδια μέρα, δηλαδή την 24η Απριλίου, μετά από ψηφοφορία των συντονιστών, με 30 ψήφους υπέρ και 26 κατά, αποφασίσαμε να μπει στη διαέρηση αδιάταξη το θέμα της Επιτροπής μας. Το θέμα δηλαδή εννοώ των παρανόμων δραστηριοτήτων και πρακτικών στη Βουλγαρία κατά πολιτικών επιχειρηματιών και δημοσιογράφων. Το ΕΛΚ όμως διαμαρτυρήθηκε και ζήτησε να γίνει ψηφοφορία από την πλήρη Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 192 του κανονισμού, γι' αυτό και ψηφίζουμε σήμερα. Τα καταλάβατε? Όχι. Α, καταλάβατε. Λοιπόν, ορίστε κυρία Ματθεού. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, Γεια σας παρακαλώ να σέβεστε τους συναδέλφους που μιλούν. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να σας πω ότι το ΕΛΚ δεν διαμαρτυρήθηκε για την ψηφοφορία 26 με 30, αλλά όπως ξέρετε από τους συντονιστές πρέπει να υπάρχει μεγάλη πλειοψηφία για κάθε απόφαση και γι' αυτό ζητήσαμε να γίνει η σημερινή. Αλλά δεν αμφισβητούμε εκείνην. Έχουμε και μία δήλωση για τη διαδικασία. Η διάσκεψη των Προέδρων θέλησε η ΕΛΕΦ να αποφασίσει εάν θα γίνει ή όχι συζήτηση εδώ. Δεν μας ζήτησαν να αποφανθούμε αν θα γίνει γενικά συζήτηση. Για τους τύπους μιλάω, για τη διαδικασία. Θα ήθελα, η ομάδα μας θα ήθελε, η Επιτροπή ΕΛΕΦ να μην υπέχει θέση δικαστηρίου. Ενώ για το θέμα αυτό μπορούμε να πούμε ότι η Κομισιόν έχει επίσημα ζητήσει να μην εξεταστεί γιατί υπάρχει προσφυγή στα δικαστήρια και η Επιτροπή Έγκλα επίσης αντιτίθεται. Και τρίτον, όπως είπατε και εσείς κύριε Πρόεδρε, η διάσκεψη των Προέδρων δεν θέλησε επίσης να παρέμβει. Και η ομάδα μας θεωρεί ότι έτσι τυπικά Υπάρχει μεν ένα θέμα, αλλά καλύτερο θα ήταν η βουλγαρική δικαιοσύνη να αποφασίσει, μάλλον παρά η Επιτροπή Ελεύ, κύριε Πρόεδρε μου. Αυτά ήθελα να πω στους συναδέλφους. Γιατί αν αρχίσουμε τώρα να εξετάζουμε όλα τα μέλη που κατά τον οποίο εκρικάζεται κάποια υπόθεση δεν θα κάνουμε πια τίποτε άλλο. Δεν είναι πολύ φρόνιμο να υποκαταστήσουμε δικαστήρια και γι' αυτό καταψηφίσαμε την, πρότα... καταψηφίσαμε την πρόταση. Μάλιστα κυρία Ματθέου, τα καταλάβαμε. Η Επιτροπή ΕΛΕΦ δεν είναι δικαστήριο. Δεν είναι δικαστήριο. Έχει όμως δικαίωμα να συζητήσει πολιτικός οποιοδήποτε θέμα που έχει πολιτικό ενδιαφέρον για την Ευρώπη ολόκληρη και όχι μόνο για τη συγκεκριμένη χώρα. Πάντως θα ψηφίσουμε. Θα ψηφίσουμε. Και έτσι θα λυθεί. Καταλάβατε ποιο παίζεται εδώ πέρα. Πρέπει να αποφασίσουμε εάν θέλουμε να συμπεριληφθεί στις συζητήσεις μας τη ΕΛΕΦ η κατάσταση στη Βουλγαρία όπως ζήτησε η διάσκεψη των Προέδρων. Έγινε ψηφοφορία από τους συντονιστάς αλλά σύμφωνα με τον κανονισμό μία πολιτική ομάδα έχει το δικαίωμα να υποβάλλει το ίδιο ερώτημα και στην πλήρη επιτροπή και αυτό θα ψηφίσουμε τώρα. Ποιοι είναι υπέρ της συμπερίληψης του θέματος αυτού για τη Βουλγαρία στις εργασίες μας. Αυτοί θα ψηφίσουν ναι. Όχι όμως αυτοί που διαφωνούν θα ψηφίσουν όχι. Λοιπόν, άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικός. Πώς υπάρχει πρόβλημα με τις κάρτες. Πάνω περισσότεροι πέντε του ΕΛΚ. Α, ναι, δεν Ναι, δεν ναι, ναι, ναι. ΕΛΚ συν πέντε λοιπόν. Συν δύο τώρα. Σοσιαλιστές συν ένας. Για να δούμε ποιος θα φύγει λοιπόν. Τώρα Τώρα εντάξει. Εντάξει. Άρχεται η ψηφοφορία. Εντάξει είναι. Πάλι ένας παραπάνω του ΕΛΚ. Ένας παραπάνω του ΕΛΚ. Ένας παραπάνω. Ποιος. «32 υπέρ 26 κατά, σχεδόν όπως, σχεδόν όπως στους συντονιστές. Εγκρίνεται δηλαδή. Εγκρίνεται τώρα έκθεση Μακοβέη. για πρόταση οδηγία Κοινοβουλίου Συμβουλίου για το πάγωμα και την κατάσχεση κερδών από εγκληματικές δραστηριότητες. Η συγγήτρια είπα η κυρία Μόνικα Μακοβέη. Η τροπολογία 163 έχει αποσυρθεί, να το ξέρετε. Αρχίζουμε λοιπόν. Έτοιμοι. Αρχίζουμε. Εμβεβαστική 6 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 70. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 71 όχι είναι ίδια με το 70 συγγνώμη 74 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 7 ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 79 ψηφ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 80 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 81 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Any problem? No. Υπάρχει κανένα πρόβλημα. Όχι, μάλιστα. 83 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 84 υπέρ, κατά. Δεν είναι σαφές. Να ελέγξουμε. Δεν είναι σαφές. Ψηφίζουμε την 84, έρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Το ΕΛΚΑ ψηφίζει με έναν παραπάνω, όπως και στους σοσιαλδημοκράτες. Να βγει ένας, παρακαλώ. Και από τη μία και από την άλλη ομάδα. Ωραία. Λοιπόν, τι έχουμε. 29 προς 24 εγκρίνεται. 87 ψήφι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 90 ψήφι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 91 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 92 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 95 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 8 Α, όχι, ελέγχουμε. Ελέγχουμε την 95, εντάξει. Πηγαίνουμε πίσω στην 95, ελέγχουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Ορίστε, δεν κατάλαβα. Συγγνώμη. Τώρα άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίζουμε για την 95. Πέρας. Πάλι είναι παραπάνω από το ΕΛΚ. Ένας παραπάνω. Εντάξει τώρα είμαστε. 23 προς 31. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 8. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Προφορική 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 9. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεν δεν εγκρίνεται. Συμβαστική 9. Εγκρίνεται. Λοιπόν, πού πάμε τώρα. Στην 109. Ψήφι υπέρ. Κατά. Δεν είναι σαφές. Ελέγχουμε την 109. Ψηφίζουμε. Πέρας φοφορίας 14 υπέρ 42 κατά. 111. 111 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 112 ψήφι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 116 υπέρ, όχι, 113 με συγχωρείτε, 113 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 116 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 117 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 119 υπέρ, κατά εγκρίνεται 118 υπέρ κατά απορρίπτεται 121 υπέρ κατά εγκρίνεται 123 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 124 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 126 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 127 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 128 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 130 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 131 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 134 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 133 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 135 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 136 να ελέγξουμε την 135. Ελέγχουμε την 135. Now closed. Πέρας ψηφοφορίας. Ένας από το ΕΛ παραπάνω. ...30 προς 27... ...εγκρίνεται... ...λυπούμε. Πάμε στην 25 υπέρ κατά αποχές νομίζω έχουμε τον εισηγητισμό ψήφων με πριν άρα μάλλον εγκρίνεται 138 138 όχι 26 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 141 υπέρ. Κατά απόχέ, εγκρίνεται. 142 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 144 υπέρ. Κατά αποχέ απορρίπτεται. 143 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 145 υπέρ. Κατά αποχές Απορρίπτεται. Όχι. Ελέγχουμε. Αλλά να σκόνετε τα χέρια σας αλλιώς. 147. Συγγνώμη. 147. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Ένας παραπάνω από το ΕΛΚ. 24 29 απορρίπτεται. 145 λέει τώρα. Απορρίπτεται. 147 υπέρ. Against. Κατά. Οι σοσιαλιστές. 147. 147. What do we... 147. Ψήφι υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίπτεται.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 κατά αποχές απορρίπτεται 154 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι απορρίπτεται αλλά επειδή δεν είναι σαφές να ελέγξουμε είναι 154 άρχεται η ψηφοφορία πέρας 32 προς 24 εγκρίνεται λοιπόν 155 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 156 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 29 υπέρ. Όχι, 157. 157. Την προσπέρασα υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται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 Όχι, όχι. Έκλεισε. Τρει. Τρεις αποχές. Yes. Just, I just want to thank you very much to all my... Θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες μου προς όλους του συναδέλφους οι οποίοι συνεισέφεραν στην έκθεση, η κυρία Μακοβέη. Πρώτα σας ευχαριστώ πολύ, αλλά δεν έχουμε ολοκληρώσει. Έχουμε άλλη μία ψηφοφορία κάπως έτσι ιδιαίτερη για την Επιστημονική Επιτροπή του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, ΦΡΑ. Ακούσαμε το πρωί τον ε, Διευθυντή, τον κύριο Μόρτιν Τζέρν. Ψηφίζουμε τώρα λοιπόν τους υποψηφίους. Έχουμε ένα κατάλογο για μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής Ο καθένας από εσάς μπορεί να ψηφίσει το πολύ 11, το πολύ 11 μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής. Λοιπόν, θα προχωρήσουμε ως εξής. Θα αναγνώσω και τα 21 ονόματα των εμπειρογνωμόνων οι οποίοι επελέγησαν για τον κλειστό κατάλογο, τον κατάλογο προεπιλογής και θα ψηφίσουμε ξεχωριστά τον καθένα. Εσείς, επαναλαμβάνω, μπορείτε να ψηφίσετε μέχρι το πολύ 11. Δηλαδή 11 φορές το πολύ μπορείτε να ψηφίσετε. Αυτοί οι οποίοι θα καταταγούν σε αυτό τον πίνακα υψηλότερα θα είναι αυτοί φυσικά που θα έχουν συγκεντρώσει τις περισσότερες ψήφους. και θα φτιάξουμε λοιπόν ε, τον πίνακα των ε, έως και 11 υποψηφίων που θα έχουν πάρει τις περισσότερες ψήφους. Παραλαμβάνω πρώτα ψηφίστε ηλεκτρονικά μέχρι και 11. Να σας πενθυμίσω κάτι ακόμα. Η σημερινή Επιστημονική Επιτροπή του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων η θητεία της λίγη στις 3 Ιουνίου του 2013. Σε ό,τι αφορά το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού, υπάρχει μια διάταξη, η οποία προβλέπει ότι το εν λόγω σώμα, ο οργανισμός δηλαδή θεμελιωδών δικαιωμάτων και συγκεκριμένα το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να συμβουλευτεί το Κοινοβούλιο πριν ορίσει τα 11 ε, μέλη που θα παρτίζουν την Επιστημονική Επιτροπή. Έχουμε λοιπόν αυτό το κατάλογο προεπιλογής με τους 21 επιλέξιμους υποψηφίους και πρέπει να την εγκρίνουμε την ε, λίστα αυτή με το σύστημα που σας προανέφερα. Δεν μπορείτε βέβαια ούτε να ψηφίσετε κατά ούτε να απόσχετε έτσι. Δεν υπάρχει αυτό. Είναι λίγο διαφορετική από τις άλλες ψηφοφορίες, δεν είναι και τόσο δύσκολη όμως παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, έχουμε ένα ελάχιστο αριθμό. Πρόεδρος, όχι. Απλά εμείς θα κατατάξουμε τους υποψηφίους ανάλογα με τις ψήφους που θα συγκεντρώσει ο καθένας. Και ο ανώτατος αριθμός τους θα είναι 11. Κατώτατο δεν υπάρχει, λέει ο κύριος Μέλο, όχι. Μπορείτε να ψηφίσετε όσε φορέ από 0 έως 11. Okay. Είναι μυστική η ψηφοφορία. Λοιπόν, ηλεκτρονικά θα ψηφίζουμε. Και το μηχάνημα θα κάνει τη δουλειά. Λοιπόν, θα του κατατάξουμε. Παναλαμβάνω, η πρώτη 11. Ψηφίζουμε λοιπόν. Έχετε αλφαβητικά τους υποψηφίους. Ξεκινάμε λοιπόν με την Rosemary μπερν. Ψηφίζουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Φυσικά δεν θα ανακοινώσουμε το αποτέλεσμα τώρα, στο τέλος. Second. Δεύτερο όνομα. Ολιβιέ Ντε Σιουτέρ. Ψηφίζουμε, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Τρίτος υποψήφιος Χαν Έντσιγκερ. Κύριε Ζόμερ. Κοίταξτε, έχω μία ερώτηση για την ε, ψηφοφορία. Αν ε, δεν θέλω να υπερψηφίσω κάτι, πρέπει να ψηφίσω με όχι ή να απέχω. Γιατί αν απέχω, τότε καταπίπτει η ε, μυστική ψηφοφορία. Γιατί από τη στιγμή που ψήφισα, ψήφισα ναι. Μήπως μπορείτε να μου εξηγήσετε τι συμβαίνει. Όχι. Ούτε όχι, ούτε αποχή. Ναι, αλλά άμα είναι έτσι, ε, τότε δεν υπάρχει πλέον μυστική ψηφοφορία. Σωστό αυτό που λέτε, δίκιο έχετε σε αυτό. Τι να πω. Yes, Frau Holmeier. Herr Vorsitzender. Κύριε Πρόεδρε, αν θέλετε μυστική ψηφοφορία τότε είναι αδύνατον να ψηφίζει κανείς μόνο ναι. Γιατί όλοι βλέπουν τι ψήφισαν οι διπλανοί. Είτε λοιπόν θα ψηφίζουμε και με όχι, γιατί είναι χαζό να έχουμε μυστική ψηφοφορία όπου όλοι βλέπουν τι ψηφίζουμε. Δηλαδή από τη στιγμή που ψηφίζω είναι σαφές ότι ψηφίζω ναι. Όλη αυτή η διαδικασία εντάξει είναι απαράδεικτη. Not the names are recollected. The names, the names of members voting are not recollected by the system. It's an electronic secret ballot. No, just, just let me. I mean, we shouldn't, we shouldn't be interrupting because we are. Λοιπόν, δεν θα έπρεπε να διακόπτουμε γιατί είμαστε εν μέσω ψηφοφορίας. Θα σας εξηγήσω όμως. Το προείπα. Είναι ιδιαίτερη η ψηφοφορία αυτή και το σύστημα είναι ιδιαίτερο. Είναι μυστική η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρα ε, δεν μπορεί να ξέρει κανείς ποιος ψηφίζει υπέρ με αυτό το ηλεκτρονικό σύστημα. Δεν μπορεί κανείς να ψηφίσει κατά ή να απόσχει. Απλά ψηφίζουμε υπέρ των υποψηφίων, όποιον θέλουμε. Και μπορείτε να ψηφίσετε μέχρι 11 ο καθένας σας.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 ψηφίζουμε ναι, λέτε ότι άπαξ και πατάει κάποιο το κουμπί, ξέρουμε ότι ψηφίζει υπέρ κάποιου ψηφίζει. Α, τώρα το κατάλαβα. Άρα, τι να κάνουμε, α βάλουμε και την αποχή. Υπάρχει και δεύτερη επιλογή, άρα μπορείτε να πατήσετε είτε αποχή είτε υπέρ. Άρα θα πατάτε όλοι ένα κουμπί και δεν θα ξέρει κανεί τι πατάτε. Πατάτε πράσινο, πατάτε λευκό, εσείς θα το ξέρετε στην καρδιά σας μέσα. Λοιπόν, άρα ψηφίζετε είτε υπέρ είτε αποχή. Μέχρι 11 μπορείτε να ψηφίσετε. Αλλιώς πατάτε το μεσαίο κουμπί. Αποχή. Άρα μπορείτε να ψηφίσετε είτε υπέρ είτε αποχή. Που βέβαια δεν θα καταμετρηθεί από το μηχάνημα. Οι αποχές δεν θα καταμετρώνται. Λοιπόν, έτσι θα προχωρήσουμε, έτσι. Τι κάνουμε. Να ξαναρχίσουμε. Εντάξει, ξαναρχίζουμε. Από την αρχή. Λοιπόν, πάμε πίσω. Ξεκινάμε με την Rosemary Byrne. Άρχεται η ψηφοφορία. Rosemary Byrne. Πέρασε. Ολιβιέντε Σιτέρ. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Αν Έντσιγκερ. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Πάτρικ Φέστη. Άρχεται η Πέρας. Ροσέ Μανουέλ Φρέσνο, άρχη του σχολείου. Πέρας. Μάρτιν Γραμμάτικοφ, άρχεται ψηφοφορία. Γραμμάτικοφ. Πέρασε. Κωνσταντς Γκρέβε, κάπως έτσι. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Κλάος Κρίστιαν Γκούλμαν. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Κριστίν Κρούμα. Άρχεται ψηφοφορία. Ζώσεφ Μάρκο. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Γιωχάννα Νιέμι. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Πάμε στο νούμερο 12. Μάικλ Κορνίλιους Φλάχερτη. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. 13. Σέι Νίλ ο Χίγγινς. Άρχεται η ψηφοφορία. 4 Gerard Quinn άρχεται η ψηφοφορία πέρασε Δεκαπέντε Αναμαρία Σαλίνας Δεφρίας άρχεται η ψηφοφορία Ταρσής. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Το 17. Χάνες Τρέτερ. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 18. Φρανσουάς Τιλικένης. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. 19. Δεκαεννέα. Κριστίνα Βαντέρκιν Άρχεται ψηφοφορία. Πέρασε ψηφοφορίας 20 Ρόμαν Βιερουζεύσκη. Άρχεται Και λίγη ψηφοφορία. 21. Τζον Ρέντς, άρχιτε ψηφοφορία. Και λίγη. Σας ευχαριστώ όλους. Σας ευχαριστώ όλους, σας ευχαριστώ όλους. Μια αναγγελία. Πριν περάσουμε στο επόμενο σημείο τη μερικής διάταξη. μου ζητήθηκε να σα υπενθυμίσω ότι αυτή τη στιγμή, ταυτόχρονα δηλαδή, δίπλα συνεδριάζει στο 4Q2 η Επιτροπή ΚΡΙΜ. Πολλά μέλη τη επιτροπή Λίμπε είναι μέλη και τη επιτροπή ΚΡΙΜ. υπάρχει μια διακοινοβουλευτική συνεδρία με τα Εθνικά Κοινοβούλια για το θέμα ρόλος και εμπειρίες των Εθνικών Κοινοβουλίων στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, της διαφθοράς και του ξεπλήματος χρήματος. Προς ενημέρωσή σας, στην ημερήσια διάταξη του ΚΡΙΜ, της Επιτροπής ΚΡΙΜ, για το οργανωμένο έγκλημα, τη διαφθορά και το ξέπλυμα χρήματος, η συζήτηση θα γίνει παρουσία του εισηγητού κυρίου Γιακολίνο στις 4 παρα 10 θα ξεκινήσει και για τα τρία αυτά θέματα. Πάμε στο επόμενο σημείο της μερισιάς διάταξης. Moving on, please, those leaving the room. Παρακαλώ. Ησύχως όσοι θέλουν να αποχωρήσουν. Και παρακαλώ να έχω την προσοχή σας για το επόμενο σημείο. Αφορά τη Συρία. Αποστολή αντιπροσωπείας για τους Σύρους πρόσφυγες στην Ιορδανία. Είναι το σημείο 16. Παρακαλώ. Την προσοχή σας παρακαλώ. Ησυχία. Ησυχία στην αίθουσα παρακαλώ. Πίσω εκεί ηρεμία. Λοιπόν, σημείο 16, αποστολή αντιπροσωπείας για τους Σύρους πρόσφυγες στην Ιορδανία. 11 με 14 Φεβρουαρίου έλαβε χώρα αυτή η επίσκεψη. Ουσιαστικά θα γίνει η παρουσίαση της έκθεσης της αντιπροσωπείας και θα συζητήσουμε με την Επιτροπή και την Υπατή Αρμοστία των Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες. Και για το, με το Διεθνές Γραφείο Μετανάστευσης, ο κ. παπα Παρακαλώ ησυχία, λέει ο πρόεδρο. Και όσο Πανικολάου. Κύριε Πρόεδρε, στην μέση διάταξη το θέμα αυτό προβλέπεται να συζητηθεί από τι 4 και 10 και μετά. Αν είναι δυνατόν λοιπόν θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα ώστε ο εισηγητή και οι σκιώδει να έλθουν. Ο κύριο Πύρκα για παράδειγμα δεν είναι εδώ. Ενώ αυτοί που ήταν μέλη τη αντιπροσωπείας, αυτό, αυτό εννοούσα. Διάλειμμα λοιπόν 20 λεπτών γιατί υπάρχουν ορισμένοι που θέλουν να είναι σε αυτό το σημείο και προβλεπόταν στις 4 και 10 να ξεκινήσει η συζήτηση άρα δεν είναι εδώ ακόμη. Κάνουμε διάλειμμα μέχρι τις 4 και 10.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 Please, we may have your attention. We're getting restarted. We'll resume our work, okay? As I said, this is the point concerning the... Λοιπόν, τώρα το θέμα για την αποστολή μας στη Συρία και τους πρόσφυγες από την Ιορδανία, α, στην Ιορδανία. Το Φεβρουάριο έγινε. Όπως ίσως θυμάστε, τέσσερις ήταν στην αντιπροσωπεία. Μεταξύ των οποίων Αργεντίνη, Μπίρκοφ, η Γιάννης Μαρινέσκου και ο ίδιος. I will, I will uh, Θα σας πω σύντομα ποιες είναι οι εντυπώσεις μας. Έχουν συνοψιστεί και γραπτός και διανυμηθεί. Ήταν πολύ συγκινητική η εμπειρία. Uh, checking mostly, uh... Κυρίως θελήσαμε να δούμε ποια είναι η κατάσταση των προσφύγων από τη Συρία στην Ιορδανία. Και επισκεφθήκαμε το στρατόπεδο Τσάτρι. Θα θυμάστε ότι το 11 άρχισε το πρόβλημα. 4 εκατομμύρια περίπου. Εκτοπίστηκαν, μετατέθηκαν και 2 εκατομμύρια σύμφωνα με την ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ πάνω από τους μισούς στην Ιορδανία, το Λίβανο, το Ιράκ και την Τουρκία είναι παιδιά και το 40% κάτω της ηλικίας των 11 μικρά παιδιά λοιπόν σχεδόν 90% των προσφύγων έφτασαν στην Ιορδανία το 11. Η Ιορδανία λοιπόν είχε τεράστιο αριθμό προσφύγων που έρχονταν εκεί και ο Ισήρη στην Ιορδανία είναι τώρα περίπου 200.000 ή 250.000 εγγεγραμμένοι πρόσφυγες. Η επίσκεψη στο στρατόπεδο Σάντρι χρειάστηκε ολόκληρη μέρα. Σχεδόν 100.000 ζουν εκεί σε ένα στρατόπεδο που δεν υπήρχε καν πριν από μερικά χρόνια. Κατασκευάστηκε τον Ιούλιο του 11. Είναι πολύ μεγάλη η συγκέντρωση ανθρώπων εκεί, η πυκνότητα. Τους βοηθάνε ορισμένες μη κοιμητικές οργανώσεις, η UNICEF, η ΥΠΑΤΗ Αρμοστία, IOM και THW, καθώς και το Save the Children. Βέβαια υπάρχει θέμα ασφαλείας εκεί γίνονται γάμοι ανηλίκων, λαθρεμπόριο, χρήση ναρκωτικών, πετροπόλεμοι. Εκτός από αυτό το στρατόπεδο όμως υπάρχουν και πολλοί πρόσφυγες στις πόλεις γιατί 80% των σύρων προσφύγων ζουν στις πόλεις και αυτό επηρεάζει αρνητικά τις υποδομές, την υγεία, τις κοινωνικές υπηρεσίες κλπ. Πιέζεται πολύ λοιπόν η Ορδανία για να αντιμετωπίσει αυτά τα προβλήματα. Επίσης επισκεφθήκαμε κέντρα καταγραφής προσφύγων, σύνορα, οριακά φυλάκια συναντήσαμε υψηλόβαθμους υπαλλήλου των Συριακών Υπηρεσιών, του Υπουργείου Εξωτερικών, του Υπουργείου Σχεδιασμού και του Υπουργείου Εσωτερικών. Συγκεκριμένα, τον Υπουργό, ο Υπουργός Εξωτερικών μας τόνισε ότι η Ορδανία έχει πολιτική ανοιχτών φυρών και δεν εκδίδει τους πρόσφυγες. Ο Υπουργός Εσωτερικών τόνισε ότι χρειάζονται πολύ περισσότεροι πόροι για να διατηρηθεί η ασφάλεια και η κοινωνική περίθαλψη, ιδίως για τις γυναίκες και τα παιδιά. Και βέβαια ο προπολογισμό που διατίθεται από την Ιορδανία δεν επαρκεί. Τονίζουν λοιπόν την ανάγκη που χρειάζεται για περισσότερη συνεργασία της διεθνούς, με τη διεθνή κοινότητα και φυσικά και από την Ευρώπη. Συναντήσαμε και εκπροσώπους μη κυβερνητικών οργανώσεων και τελικά γράψαμε τα συμπεράσματά μας όπου εκφράζαμε την ανησυχία μας για την ανθρωπιστική κρίση εκεί και εκτιμήσαμε δεόντως τις προσπάθειες της Ιορδανίας και της διεθνούς κοινότητας για να βοηθήσει την Ιορδανία. Παρατηρήσαμε όμως ότι οι δυνατότητες της είναι σχεδόν, έχουν σχεδόν εξαντληθεί και υπάρχουν λίγοι πόροι Ούτε η στήριξη της διεθνούς κοινότητας δεν αρκεί για να αντιμετωπίσει τις βασικές ανάγκες των προσφύγων. Τονίσαμε λοιπόν την ευθύνη που έχει η διεθνής κοινότητα. Ζητήσαμε από τις Ιορδανικές αρχές να διατηρήσουν ανοιχτά τα σύνορα και είπαμε ότι θα έπρεπε να βοηθήσουν και οι γειτονικέ αραβικές χώρες για τη διευθέτηση και αντιμετώπιση της κρίσης και μακροπρόθεσμα θεωρούμε ότι ένα περιφερειακό πρόγραμμα προστασίας είναι απαραίτητο για να υπάρξει μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων εκεί και παραγόντων όπως μήκη όμικρον συνοριακών φυλάκων ζητήσαμε συγκέντρωση των προσπαθειών εκεί όπου υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη και καλέσαμε τις Ιορδανικές αρχές να διασφαλίσουν την τήρηση της τάξης εκεί και να δίνουν πρόσβαση στους, στις ανθρωπιστικές οργανώσεις εκεί κοντά στα σύνορα. Αυτή είναι λοιπόν η έκθεσή μας και προτείνω τώρα μετά την συνοπτική αυτή παρουσίαση να γίνει η συζήτηση και με τις οργανώσεις που εκπροσωπούνται εδώ στην αίθουσα. Πρώτη λέω να είναι η ύπατη αρμοστία. Ο εκπρόσωπος της είναι ο κύριος Κόχτελ, αν θέλει να μας πει τίποτε Ο κύριος Κόχτελ γυρίζει. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου δίνετε να μιλήσω για την κατάσταση στην Συρία και για την ανθρωπιστική κατάσταση στη χώρα αυτή. Πρέπει λοιπόν να παρακολουθήσουμε εκ του συνεγγύς τις εξελίξεις ε, και πρέπει ε, να αναλάβουμε τις ευθύνες μας ε, για την ε, προστασία των προσφυγών στην Ιορδανία κυρίως. Μιλάμε για 8.000 πρόσφυγες που καταφθάνουν κάθε μέρα από τις όμορες χώρες. Θέλω να υπογραμμίσω ότι η Τουρκία παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην παροχή πολύ ουσιαστικής βοήθειας. Η Τουρκία από τον Απρίλιο του 2011 έχει δεχτεί 400.000 πρόσφυγες. Άρα δηλαδή μιλάμε για περισσότερους πρόσφυγες από τους ε, ετούντες άσυλο που έχουν δεχτεί ε, όλες οι ευρωπαϊκές χώρες κατά το ίδιο χρονικό διάστημα. Είναι βέβαια δύσκολο να πει κανείς στην Τουρκία αφήστε ανοιχτά τα σύνορα με την Συρία και κλείστε τα με την, ε, την Κύπρο, τη Βουλγαρία ή την Ελλάδα. Θα ήθελα λοιπόν σήμερα να σας μιλήσω κάτι το οποίο αφορά τις ε, όλο και μεγαλύτερες ανησυχίες μας για τους Σύριους στην Ευρώπη. Είμαστε σε μια δύσκολη φάση ολοκληρώνεται το σύστημα χορήγησης ασύλου στην Ευρώπη και πρόκειται σύντομα να εφαρμοστεί το σύστημα αυτό. Πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη μας τις ε, διατάξεις που θα ε, θεσπιστούν γιατί αυτές ε, θα έχουν άμεση εφαρμογή σε αυτούς τους ανθρώπους που χρειάζονται τη διεθνή προστασία. Και πρέπει και εμείς να κάνουμε τα απαραίτητα βήματα. Ο αριθμός λοιπόν των Συρίων τον άσυλο και των προσφύγων στην Ευρώπη είναι περίπου 36.000 άνθρωποι από τον Απρίλιο του 2011. Σε πολλές χώρες ε, εφαρμόζονται ε, σωστές πρακτικές ε, που μπορούν να επενεθούν με βάση το διεθνές δίκαιο. Υπάρχουν όμως και σημαντικές ελλείψεις. Ορισμένες χώρες στέλνουν τους ετούντες άσυλο από τη Συρία σε καταβλισμούς ε, κράτησης ε, προσφύγων. Βλέπουμε επίσης ε, πολύ περιορισμένο αριθμό χορήγησης ασύλου σε πολλές χώρες και σε άλλες υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση. Οι ετούντες άσυλο πρέπει, εφόσον χρειάζονται προστασία να μπορούν να εισέλθουν στην Ευρώπη, πρέπει να έρθουν οι διατάξεις περιορισμού ε, της ε, θεώρησης και πρέπει να είναι δυνατόν οι ε, οικογένειες να επανενώνονται με ασφάλεια. Άλλα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι πρόσφυγες, στην περίπτωση αυτή οι Σύριοι πρόσφυγες, έχουν σχέση με την εφαρμογή του κατεστημένου, του κοινωνικού κατεστημένου για τη χορήγηση ασύλου η εφαρμογή γίνεται με ένα τέτοιο τρόπο που δεν, ε, δεν προβάλλονται οι ανθρωπιστικές ε, ανάγκες. Έχουν γίνει πολλά λάθη. Οι Σύριοι πρόσφυγες σε ένα κράτος μέλος ε, μπορεί να τύχουν αναγνώρισης και σε ένα άλλο κράτος μέλος να μπορούν όμως να επανωθούν πολύ εύκολα με την οικογένειά τους λόγω της συμφωνίας του Δουβλίνου. Η λύση εφαρμόζεται βέβαια με αυστηρή εφαρμογή του κοινωτικού κακεκτημένου και αυτό αμφισβητείται αν θα πρέπει να ισχύει αυτό ή να λάβουμε υπόψη μας την πραγματικότητα. Εγώ θεωρώ ότι οι αιτούντες άσυλο από την Συρία πρέπει να έχουν πρόσβαση στην Ευρώπη και εφόσον χρειάζονται να έχουν και ε, προστασία. Εξάλλου πρέπει να την χάνουν ε, τις ελάχιστες προστασίες ε, βασικών δικαιωμάτων ε, στα κράτη-μέλη, κάτι που δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Και πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα μεταφέρονται σε καταβλισμούς προσφύγων και σε κέντρα κράτησης, όπως συμβαίνει αυτό συστηματικά σε ορισμένες χώρες. Οι ετούντες άσυλο στην Ευρώπη πρέπει να αντιμετωπίζονται με τέτοιο τρόπο που ε, θα καθιστά σαφές ότι οι άνθρωποι αυτοί έχουν ε, διαφύγει και διώκονται. Ας μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και βάλωτες ε, ομάδες και αυτοί λοιπόν που φεύγουν από τη Συρία θα πρέπει να την χάνουν προστασίες, να μπορούν να ε, εγκαθίστανται στην Ευρώπη. Σε σχέση με αυτά που ανέφερα, η αρμόδια υπηρεσία έχει, έχει καλωσορίσει, χαιρετίζει την πρωτοβουλία της Γερμανίας. Ξεκινήσαμε λοιπόν τον εντοπισμό αυτών των προσφύγων ε, αρχίσαμε να εντοπίζουμε τις ανάγκες τους εγκατάστασης και στηρίζουμε εκείνα τα κράτη-μέλη που έχουν δηλώσει προθυμία να δεχτούν αυτούς τους ε, ανθρώπους ε, ε, οι χώρες αυτές προς το παρόν είναι η Σουηδία, η Δανία και η Ελβετία. Επίσης εξακολουθούμε να ελέγχουμε την κατάσταση, προετοιμαζόμαστε για το ενδεχόμενο στο μέλλον να υπάρξουν περισσότερες αιτήσει και τα κράτη-μέλη πρέπει να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν αυτές τις ανάγκες. Είναι απαραίτητο να ληφθούν βήματα να γίνουν βήματα έτσι ώστε να ε, δείξουμε την αλληλεγγύη μας με τον ε, Λίβανο, την Ιορδανία και την Τουρκία, ε, χώρες που συμπεριφέρθηκαν με μεγάλη γενεοδορία απέναντι σε πρόσφυγες που αναγκάστηκαν να φύγουν λόγω της κατάφορης παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Συρία. Και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Φρανσουά Γκέμενς που εκπροσωπεί ε, την οργάνωση ION στις ε, Βρυξέλλες. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα σας περιγράψω τις δραστηριότητες ε, του γραφείου μας στην Ιορδανία. Παρέχουμε αρρωγή ε, ως προς τη μεταφορά των προσφύγων στους καταβλισμούς. 1.500 πρόσφυγες την ημέρα εξυπηρετούνται. Ε, ξέρουμε ότι περνούν ε, τη νύχτα τα σύνορα και τους μεταφέρουμε ε, στο καταβλισμό, στο στρατόπεδο. Και έχουμε αρχίσει τώρα να τους μεταφέρουμε και στο στρατόπεδο που βρίσκεται στα Εμμυράτα. περισσότεροι Σύριοι έρχονται από την Τάχα και τα γειτονικά χωριά και στο να Νασίμπ παρατηρούνται περισσότερες διελεύσεις. Υπάρχει επίσης μια ιατρική μονάδα για τον εμβολιασμό τους ε, κατά της λαράς ε, και της πολιομιελίτιδας ε, και γενικώ δίνουμε τις απαραίτητες βιταμίνες, κάνουμε κάποιες δραστηριότητες για να ανοιχνεύσουμε ενδεχόμενα φυματίωση και έχουμε και κάποιες εκστρατείες ευαισθητοποίησης. Αυτό το οποίο έχουμε παρατηρήσει είναι και κάποια κρούσματα βίας και επιδείνωση της κατάστασης ασφαλείας στο στρατόπεδο και όλο και περισσότερο βιώνουμε προβλήματα με πορνεία, σεξουαλική εκμετάλλευση λόγω του τεράστιου βάρους δηλαδή πάρα πολύ μεγάλος αριθμός προσφύγων έχει συγκεντρωθεί στην Ιορδανία αυτά είχα να πω ευχαριστώ Πρόεδρος. Ωραία, τώρα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κύριος Αντουάν Λεμασόν, που είναι ο αναπληρωτής διευθυντής της Γραμματέλτα Έκονας. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε για την έκθεση όπως επίσης και για την ε, σύντομη παρουσίασή σας. Ε, όλα αυτά είναι πολύ ενδιαφέροντα γιατί αν συγκρίνουμε τον αριθμό των προσφύγων που αναφέρονται στην έκθεση, δηλαδή 250.000 ε, καταγεγραμμένοι πρόσφυγες ε, πριν από τρει μήνες όταν επισκεφτήκατε επιτόπου την περιοχή. Σήμερα μιλάμε για 450.000. Βλέπετε λοιπόν ότι έχουμε εντυπωσιακή επιδείνωση της ε, ανθρώπινης κατάστασης. Αυτό ισχύει για την υπηρετική περιοχή της Συρίας και για τις όμορες χώρες. Τώρα έχουμε 1,4 εκατομμύρια ε, καταγεγραμμένους ε, πρόσφυγες ε, Συρίους στις όμορες χώρες. Και στις αρχές του αιτούς είχαμε 850.000. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες της κατάστασης στη Συρία που από ανθρωπιστική πλευρά η κατάσταση είναι τραγική. Εμείς πιστεύουμε ότι η σύγκρουση στη Σουρία, Συρία έχει ξεφύγει από το ανθρωπιστικό πλαίσιο. Αυτή τη στιγμή διακυβεύεται η σταθερότητα στην περιοχή, κυρίως για δύο χώρες που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα, δηλαδή το Λίβανο και την Ιορδανία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και γενικότερα η Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς την αντίδρασή τους κάναμε τα εξής. Προσπαθήσαμε να έχουμε ενεργό παρουσία επιτόπου με εμπειρογνώμονες της ΕΚΟ, στο ΑΜΑΝ, στη Βηρητό, στην Άγκυρα και στο Γκαζιαντέπ. Είχαμε ένα γραφείο στη Δαμασκό, αναγκαστήκαμε όμως ε, να το μεταφέρουμε λόγω της ε, κατάστασης ε, και βέβαια αν χρειαστεί το γραφείο αυτό μπορεί να ξανανοίξει. Έχουμε ενεργό παρουσία επιτόπου με επισκέψεις υψηλού επίπεδου. Η Επίτροπος Γεώργεβα επισκέφθηκε ήδη την Τουρκία, το Δεκέμβρη επισκέφθηκε την Ιορδανία και το Λίβανο με τον ε, είπα το αρμοστή Γκουμίτερες και θα επανέλθει στην Ιορδανία και το Λίβανο αυτή την εβδομάδα. Όπως και εσείς ε, θα επισκεφτεί ε, το συγκρότημα Ζάταρουι, θα προσπαθήσει, ε, αν το επιτρέπει η ασφάλεια, να μεταβεί στα σύνορα και στο Λίβανο θα προσπαθήσει επίσης να επισκεφτεί την Μπεκά, την κοιλάδα Μπεκά. Θα συναντηθεί με δύο πρωθυπουργού και με τους υπουργού που είναι αρμόδιοι για τους πρόσφυγες και στις δύο χώρες. με την υποστήριξη των ε, εταίρων μας, ε, των ε, ειδικών οργανώσεων των Ηνωμένων Εθνών, έχουμε καταλήξει στο ότι αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο μεγαλύτερος δωρητής. Η ανθρωπιστική βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση ανέρχεται σε περίπου 473 εκατομμύρια ευρώ. 200 εκατομμύρια έχουν ήδη εκταμιευτεί και περίπου 273 εκατομμύρια έχουν εκταμιευθεί από τα κράτη-μέλη. Τα πρώτα 273 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίσης, θέλω να πω, το ίμιση της ανθρωπιστικής βοήθειας πηγαίνει στη Συρία. Ένα τέταρτο στο Λίβανο και ένα τέταρτο της βοήθειας στην Ιορδανία. Βλέπετε λοιπόν ποιες είναι οι προτεραιότητές μας. Αφορούν αυτές τις ε, τρεις χώρες θεωρούμε ότι το Ιράκ και η Τουρκία, επειδή είμαστε αναγκασμένοι να ερχίσουμε τα προβλήματα, θεωρούμε ότι οι δύο αυτές χώρες ε, έχουν τη δυνατότητα να αντιδράσουν. Επίσης, αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να αυξήσουμε τα κονδύλια. Η Επίτροπος, ε, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής της, θα ανακοινώσει μεγαλύτερη βοήθεια. Ε, η βοήθεια θα ανέλθει σε περίπου 605 εκατομμύρια ευρώ και προσπαθούμε να προσφέρουμε ό,τι μπορούμε ε, λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση πληττεί και άλλα μέρη του κόσμου. Προσπαθούμε να έχουμε και καλύτερο συντονισμό. Ε, θέλουμε να στηρίξουμε τον Λίβανο και την Ιορδανία όπως ε, το κάνατε κι εσείς κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας. Θέλουμε να τους περάσουμε το μήνυμα να σέβονται την αρχή των ανοιχτών συνόρων. Ευχαριστούμε και εσάς που το πράξατε. Πιστεύουμε όμως επίσης τουλάχιστον από πολιτική και οικονομική σκοπιά υπολείπονται ακόμα πολλά. Αυτά που έχουν γίνει δεν αρκούν. Άρα δηλαδή είμαστε σε συζητήσεις με την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και με άλλες υπηρεσίες της Επιτροπής για να επιτύχουμε ένα περιεκτικό πακέτο που θα επιτρέψει να αντιδράσουμε αποτελεσματικά στην κρίση. Και τώρα τα σχόλια από τα μέλη. Πρώτα όμως η Κομισιόν. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Επιτροπή σας για την πρόσκληση και για τη δυνατότητα που μας δίνετε να ανταλλάξουμε απόψεις για το θέμα αυτό. Η Κομισιόν ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για την πολιτική ασφάλεια και την ανθρωπιστική κατάσταση στη Συρία και για την τύχη των προσφύγων εκεί, των προσφύγων από τη Συρία στην Ιορδανία. Ξέρουμε πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα εξαρτάσαμε την έκθεσή σας και δεχόμαστε τα συμπεράσματά της. Επίσης υποστηρίζουμε τις συστάσεις σας, αλλά θα ήθελα κύριοι βουλευτές να αναφερθώ και σε πολλές άλλες συστάσεις που έχουν ήδη γραφτεί από την Κομισιόν. Υπάρχει μία, θα χωρίσω τα πράγματα σε δύο μέρη, Πρώτον, τι γίνεται στην Ιορδανία. Δεύτερον, τι γίνεται με τους πρόσφυγες από τη Συρία στην Ένωση. Επιτόπου στη Συρία και στις γειτονικέ χώρες, καταρχήν, χορηγούμε συνεχώς ανθρωπιστική βοήθεια για τους εκτοπισμένους και τους πρόσφυγες και ή δυνατόν και στην ίδια τη Συρία μέσα. Συνεργαζόμαστε στενά με την ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ και άλλες υπηρεσίες του και η πέμπτη σας σύσταση για τη συνεχή στήριξη επειδή μεταναστευτικές, μάλλον προσφυγικές ροές συνεχίζονται και αυξάνονται πρέπει να χορηγείται βοήθεια και προστασία και ιδιαίτερα για του εκείνους που αποφάσισαν να φύγουν από τη Συρία και να καταφύγουν στις γειτονικές χώρες, Ιράκ, Λίβανο, Τουρκία, Ιορδανία. Η συνέχιση της στήριξης είναι κατά εμάς η πιο άμεση προτεραιότητα και ο συνάδελφός μου από τη Γενική Διεύθυνση ΙΚΟ είπε επίσης ότι είμαστε ακόμη, συνεχίζουμε να παραμένουμε, παραμένουμε ο κυριότερος διεθνής παράγων που χορηγεί βοήθεια εκεί. Τώρα η σημασία των γειτονικών χωρών πρέπει να κρατούν ανοιχτά τα σύνορά τους για τους πρόσφυγες από τη Συρία όπως λέτε και στη σύσταση 6. Οι χώρες αυτές που αναφέρατε, Ιράκ, Λίβανος, Ιορδανία, Τουρκία, κάνουν προσπάθειες και προσπαθεί και η Κομισιόν να σταθεροποιήσει την κατάσταση στη χώρα ώστε να υπάρχει επαρκής προστασία. Κύριε Πρόεδρε, αναφέρατε επίσης το πρόγραμμα περιφερειακής προστασίας. Παράλληλα με τις ανθρωπιστικές μας προσπάθειες, οι υπηρεσίες της Κομισιόν σε συνεχή επαφή με άλλους διεθνείς παράγοντες εφαρμόζουν ένα τέτοιο πρόγραμμα, το λεγόμενο RPP το οποίο συμπεριλαμβάνει και την Ιορδανία και το Ιράκ και το Λίβανο. Το πρόγραμμα αυτό συμφωνεί με τις τελευταίες κατευθυντήριες γραμμές της Κομισιόν για την χορήγηση ανθρωπιστικής βοήθειας, ιδιαίτερα για δράσεις υπέρ των προσφύγων. κύριος Κώσταλ από την υπα αρμοστία ανέφερε την ιδιαίτερη σημασία της Τουρκίας και γι' αυτό γίνεται μια ανάλογη προσπάθεια και για την Τουρκία από τις υπηρεσίες της Κομισιόν σε σχέση και συνεργασία με την υπα αρμοστία. Τώρα θα ήθελα επίσης να αναφέρω, ο, και αυτό νομίζω ότι είναι σημαντικό, ότι πρέπει πρέπει να έχουμε μετρημένες προσδοκίες γιατί πρέπει πρώτα να πείσουμε τις γειτονικές αυτές χώρες. Δεν μπορούμε να υπολογίζουμε σε άμεση ετοιμότητά τους για την εφαρμογή όλων αυτών των προγραμμάτων. Τέλος, έρχομαι στην κατάσταση των σύρων που ζητούν άσυλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κύριος Κοστέλ είπε λεπτομέρειες, ανέφερε λεπτομέρειες. Μέχρι τώρα οι αριθμοί ήταν χαμηλοί και διαχειρίσιμοι. 32.000 άνθρωποι έχουν, από τη Συρία έχουν ζητήσει άσυλο στην Ένωση από την αρχή της κρίσης τον Απρίλιο του 2011 και μέχρι το τέλος του 2012. 32.000. Οι τελευταίοι αριθμοί επιβεβαιώνουν περίπου 93% ρυθμό αναγνώρισης και ικανοποίηση τέτοιων ετοιμάτων από την Ένωση. Παρακαλώ σεβαστείτε το χρόνο γιατί ε, πρέπει να συζητήσουμε και για την Ουγγαρία μετά. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Φαίνεται ότι γενικά υπάρχει συνένεση μεταξύ χωρών μελών ότι οι Σύροι που προσφεύγουν στην Ένωση δεν πρέπει να εκδίδονται και να επιστρέφουν εκεί. Αλλά όπως είπε και η πατιαρμοστία σε μερικές χώρες μέλη όπως την Ελλάδα και την Κύπρο σχεδόν 0% αναγνώριση. Και εκεί θεωρείται ότι οι περισσότεροι αιτητές εσύλου που παρουσιάζονται ως Ήροι δεν είναι πράγματι. Θελήσαμε να θα συζητήσουμε αυτό το θέμα της διαφοράς των αναγνωρίσεων. Τέλος, το θέμα της επανένωσης οικογενειών. Εμείς θεωρούμε ότι τα μέλη οικογενειών σύρων που νόμιμα διαμένουν στην Ένωση πρέπει να έχουν το δικαίωμα της οικογενειακής επανένωσης και ζητήσαμε από τα κράτη-μέλη να επιδείξουν γενεοδορία στη χορήγηση θεωρήσεων. Επίσης, η σύγκληση των προσπαθειών μεταξύ χωρών μελών συζητήθηκε επίσης τον Μάρτιο Λυπούμε που μακρηγόρησα, αλλά ήθελα να σας τα πω όλα. Τώρα λοιπόν ε, ε, τα μέλη που συμμετείχαν την προσωπή έχουν το λόγο. Κύριος Πίλκα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, πρέπει να πω όλα αυτά που ακούσαμε ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα, όπως και το έγγραφο της Επιτροπής που το μελέτησα. Επιτρέψτε μου να αναφερθώ σύντομα στην επίσκεψή μας που έδειξε ένα πράγμα ότι στην Ιορδανία οι Ιορδανικές οργανώσεις κάνουν θαυμάσια δουλειά και οι υπόλοιπες οργανώσεις, οι διεθνείς οργανώσεις, ο IOM εκπροσωπείται εδώ και αυτοί εργάζονται θαυμάσια. Ε, συνεργάζονται όλοι αυτοί οι φορείς ε, και εκεί όπου είναι σωστή η συνεργασία, είναι πάρα πολύ καλή και η βοήθεια που προσφέρεται. Η δεύτερη παρατηρήση που θέλω να κάνω είναι η εξή. Μετά από πολλές συζητήσεις με τους πρόσφυγες, αποδείχτηκε ότι ο απότερος στόχος είναι πρόθεσμα εκτός χώρας ίσως και μέσα στη χώρα να αποκτήσουν οι πρόσφυγες ασφάλεια για να επανέλθουν το συντομότερο δυνατόν. Οι ίδιοι πρόσφυγες είπαν ότι κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στους καταβλισμούς πολλές φορές επισκέπτονται τα σπίτια τους για να δουν πώς είναι τα πράγματα, μήπως ε, έχουν ε, προκύψει λαιλασίες και παρεμφερεί. Αυτό λοιπόν σημαίνει όπως ε, αναφέρει και η Επιτροπή στο εγγραφό της, ε, η προτεραιότητα είναι να παρέχεται βοήθεια επιτόπου έτσι ώστε αυτή να ε, συνεπάγεται ουσιαστικά ασφάλεια και η ασφάλεια δίνει το αίσθημα στους ανθρώπους ότι μπορούν από αυτούς τους παραμεθόριους καταβλισμούς να επιστρέψουν στη γενέτειρά τους. Πρέπει λοιπόν να παρέχετε βοήθεια γιατί οι ε, γειτονικές χώρες και αυτό θέλω να το υπογραμμίσω οι όμορες χώρες είναι εκείνες που κατά κύριο λόγο μπορούν να προσφέρουν την, την καλύτερη βοήθεια. Γιατί ε, όσοι πάνε σε αυτές τις γειτονικέ χώρες μπορούν πολύ πιο εύκολα να επιστρέψουν. Εξάλλου θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι ε, το των δυνατόν ε, στους μεγάλους καταβλησμούς πρέπει να υπάρχει εφταξία. Γιατί μιλάμε για μικρές πόλεις κατ' ουσίαν, οι οποίες ε, όμως πολλές φορές χαρακτηρίζονται από παντελή ανομία και έτσι λοιπόν στους καταβλισμούς αυτούς εμφανίζεται όλο και περισσότερο εγκληματικότητα, εκμετάλλευση, πορνεία. Και εμείς αυτά τα διαπιστώσαμε επιτόπου, άρα δηλαδή πρέπει να βοηθήσουμε. Να βοηθήσουμε έτσι ώστε στους καταβλισμούς να ε, διασφαλίζεται η εφταξία. Εμείς ε, μιλήσαμε με την ε, αστυνομία της Ιορδανίας, τους είπαμε να είναι παρόντες επιτόπου για να λειτουργούν αποτρεπτικά. Νομίζω ότι αυτά είναι τα δύο βασικά σημεία στα οποία πρέπει βραχυπρόθεσμα να εστιάσουμε την προσοχή μας. Ε, αντίθετα, ε, το όλο θέμα των ε, νέων οικισμών αυτό δεν συζητήθηκε γιατί δεν το επιθυμούν οι πρόσφυγες οι, πρό... οι πρόσφυγες επιθυμούν ε, να βοηθηθούν ε, στα σύνορα, τόπου εκεί που βρίσκονται και αυτό πρέπει να στηρίξουμε γιατί μόνο αυτό το κρίνουμε παραγωγικό. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Ρισπέκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομη. Έχω πάει ε, στις αρχές αυτήν πέρυσι ε, στην περιοχή και οι διαπιστώσεις που περιγράφεται στην έκθεση, ε, στην αναφορά της αντιπροσωπείας, δεν τη διάβασα βέβαια γιατί πριν από λίγο την πήρα, επιβεβαιώνουν πάντως ε, την καταστροφική από ανθρωπιστικής, για να μην πω απλά ανθρώπινης πλευράς κατάσταση στην οποία ε, διαπιστώνουμε ότι ισχύει. Και επίσης βλέπουμε να υπάρχει και μια πολιτική αδυναμία, ιδίω από την πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία δεν μπορεί να δώσει απαντήσει σε ό,τι αφορά την προστασία των προσφύγων. Για να ε, αντιμετωπίσει αυτά τα προβλήματα που βλέπουμε. Σχεδόν να ε, εξαφανίζεται κάτω από την μπροστά στα μάτια μας ένας ολόκληρος πολιτισμός. Εκατομμύρια είναι οι νεκροί. Είμαστε ο πρώτος ε, χρηματοδότης, ο πρώτος δερτής, αλλά πρέπει να δώσουμε μια γρήγορη απάντηση. Έχουμε τις μη κυβερνικές οργανώσεις, ανθρωπιστικές οργανώσεις, οποίες πρέπει να βοηθήσουμε ή, πρέπει να προωθήσουμε την ε, πιστιστική βοήθεια στη Συρία. Δεν ξέρω, θα μας πείτε εσείς αν έχετε απαντήσεις. Φαίνεται ότι η πιστητική βοήθεια, και λέω φαίνεται, εσείς θα μας πείτε, ότι ε, δεν φτάνει στους αποδέκτες που πρέπει. Δεν την ε, παίρνουν αυτή τη βοήθεια αυτοί που την έχουν ανάγκη, αλλά πηγαίνει ε, στον Πασάρ Αλσάραφ και ότι ε, Λάσαντ και ο πληθυσμός που υποφέρει, όποιοι έχουν κάποιες χρόνιες παθήσεις, ε, είναι καταλελειμμένοι εντελώ στην τύχη τους. Ναι, μεν είμαστε οι πρώτοι χρηματοδότες, οι πρώτοι αλλά ποια είναι η κατάσταση στην πράξη σε σχέση με την παροχή βοήθεια τελικά. Δεν μπορούμε να μετρήσουμε τα αποτελέσματα. Τώρα, η δεύτερη πτυχή, ε, το δεύτερο σκέλος παρουσιάστηκε πάρα πολύ καλά για τους ε, ετούντες άσυλο ε, στην Σουηδία που ήμουν πριν από τρεις ημέρες και χάρη στη Συριακή κοινότητα εκεί που είναι πολύ άριθμη είναι χιλιάδες οι Σύριοι ε, οικογένειες ε, Συριακές οι οποίοι χαίρουν προστασία εκεί. Επειδή υπόθηκε και πριν ότι θα πρέπει να υπάρχει αλληλεγγύη και ίσως να είναι πιο ελαστική ε, η όρη για την παροχή ασύλου επειδή βλέπουμε την απάνθρωπη κατάσταση που επικρατεί εκεί γιατί δεν μπορούμε να το παραγνωρίζουμε σήμερα. Υπάρχουν πολιτικές πτυχές, ε, από χθες συζητούμε το θέμα της χρήσης ημίχημικών. Ποιο θέλει τα χημικά όπλα, είναι όλη η συζήτηση εκεί επικεντρωμένη και δεν στηρίζουμε αυτόν τον λαό, τον μαρτυρικό αυτό λαό που είναι πράγματι ένας λαός που υποφέρει. Τώρα σας ευχαριστώ πολύ κύριε Ρισπέκ και όλους εσάς που πήρατε το λόγο θέλω να σας ευχαριστήσω. Δεν βλέπω να έχει σηκώσει κανείς το χέρι του να ευχαριστήσω για την παρουσίαση αυτή της έκθεσης της αντιπροσωπείας για τους Σύρους πρόσφυγες στην Ιορδανία. Παρακαλώ. Κύριε Εγώ αυτό που θέλω να ξέρω είναι αν ε, η βοήθεια επιστηστική που στέλνετε, ε, στέλνετε για τους Σύρους πρόσφυγες, εάν ε, τελικά φτάνει ή δεν φτάνει στους αποδέκτες. Μήπως πηγαίνει στο Μπασάρα Τελικά αυτό αληθεύει δεν αληθεύει. Είναι συγκεκριμένη ερώτηση λέει ο Πρόεδρος. Ο εκπρόσωπος της Αρμοστίας, Κοστέλ, μήπως θα ήθελε να απαντήσει για να περάσουμε μετά στο επόμενο σημείο, το γκρικό ζήτημα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, θα απαντήσω στη μετρική μου γλώσσα. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για την διανομή τροφίμων στην Συρία, αλλά συνεργαζόμαστε με το Παγκόσμιο Πιστιστικό Πρόγραμμα και πολλές κυβερνητικές και μη κυβερνητικές οργανώσεις για να παράσχουμε βοήθεια εκεί που υπάρχει ανάγκη στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση ή από την αντιπολίτευση ε, ζώνη. Τώρα το να σας πω ότι ε, δεν υπάρχει κανένα τέτοιο κρούσμα, ούτε είναι αλήθεια αυτό, ούτε και αλήθεια είναι ότι γίνεται και συστηματικά. Από το Μάρτιο, για να πάει κανεί από, το, από τη Δαμασκό στο Χαλέπι, υπήρχαν 32 ε, σημεία ελέγχου. Λίγα, ε, ήταν στα χέρια ε, της κυβέρνησης ε, και από τα άλλα ε, τα μισά σχεδόν είναι σε χέρια Τσετσένων και άλλων. Δηλαδή είναι ότι είναι κάση Σύρους. Είναι δύσκολο να εργαστεί κανείς στη Σύρια. Αυτό θέλω να πω. Αυτά γίνονταν στις αρχές Μαρτίου. Τώρα από τη Δαμασκή που κανείς στο Χαλέπ σήμερα έχει πολύ λιγότερα πολύ περισσότερα σημεία. Είναι πιο πολύπλοκη η κατάσταση τώρα, είναι ρευστά τα πράγματα, δεν είναι ξεκάθαρα. Σήμερα μπορεί ε, να ελέγχει κάποιο σταθμό η αντιπολίτευση ε, και την άλλη μέρα η ε, κρατική. Και υπάρχουν δυσκολίες. Είναι δύσκολο να φτάσει βοήθεια σε αυτούς που τη χρειάζονται, στον πληθυσμό δηλαδή που τη χρειάζεται. αυτά προς το παρόν λοιπόν. για την ε, κατάσταση των σύρων προσφύγων στην Ιορδανία και περνάμε στο επόμενο σημείο. Στο σημείο υπερτμών 10... Στο σημείο υπαρτμών 17. Εδώ θα εξετάσουμε το σχέδιο της έκθεσης ε, που έχει καταθέσει ο συνάδελφός μας ο κύριος ε, Ταβάρης. Στις 12 ε, Φεβρουαρίου του 2012 είχαμε ένα ψήφισμα για τις πολιτικές εξελίξεις στην Ουγγαρία και έχουμε την εντολή να παρακολουθήσουμε την κατάσταση. Κατά πόσον δηλαδή έχουν ε, γίνει δεκτές και σεβαστές οι απόψεις μας και ε, ποια είναι η απόψή μας. Ο κύριος Ταβάρες ε, έχει παρουσιάσει έγγραφα εργασίας και τώρα θα καταθέσει το σχέδιο της έκθεσής του. Κύριε Ταβάρες, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, Μπροστά μας έχουμε πολλή δουλειά όσον αφορά τα έγγραφα εργασίας ε, τα οποία προετοιμάσαμε. Και πολλά από αυτά έχουν ε, υπογραφεί και από τις πολιτικές ομάδες, από τους ε, σκιώδεις συγητές. Πήγαμε στη Βουδαπέστη και είχαμε ουσιαστικές συζητήσεις με τις αρχές της Ουγγαρίας Τώρα λοιπόν καταλήξαμε σε μία φάση όπου όλες οι πολιτικές ομάδες συμφωνούν με το έγγραφο. Τα σχόλια τα έχουμε συμπεριλάβει στο έγγραφο εργασίας και ακολουθήσαμε μια συγκεκριμένη μέθοδο την οποία και θα σας ε, εξηγήσω. Καταλήξαμε τελικά στο σχέδιο έκθεσης. Ας ξεκινήσουμε Ας ξεκινήσουμε με ένα ποίημα ενός Ούγκρου ποιητή του Πέτο Σάντορ, ίσως και το σημαντικότερο, της Επανάστασης του 48. Το ποίημά του λοιπόν, ελπίζω να τα καταφέρω στα ουγγρικά, που σημαίνει κατά προσέγγιση δεν υπάρχει πατρίδα, δεν υπάρχει σπίτι, στία όπου δεν υπάρχουν δικαιώματα. Αυτό λοιπόν το απόσπασμα κατ' ουσίαν δείχνει το τι χρωστά η Ευρώπη στην πλούσια ουγγρική ιστορία. Δεν υπάρχει όμως στην έκθεσή μας για αυτό το λόγο, αλλά διότι επιθυμούμε να δείξουμε ότι αν δεν έχει κανείς πατρίδα δεν αισθάνεται ασφαλής και αυτό ισχύει όταν ε, δεν ε, έχει κανείς δικαιώματα ή όταν δεν γίνονται σεβαστά τα δικαιώματά του. Κατόπιν τούτου μπορεί κανείς επίσης να ισχυριστεί ότι εκεί όπου ε, κάνουμε βήματα στο να εγγυηθούμε δικαιώματα αυτό συνεπάγεται ότι κατασκευάζουμε και στίες Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να ανεγείρουμε ένα σπίτι δημοκρατικών δικαιωμάτων, τάξης ε, κράτους δικαίου για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες, για όλα τα κράτη-μέλη. Αν δούμε λιγάκι τις συνθήκες, το πρώτο και σημαντικό που διαβάζουμε είναι στο άρθρο 2. Το άρθρο 1 λέει ότι τα κράτη-μέλη επιθυμούν να ιδρύσουν ένωση. Το άρθρο 2 αναφέρει ότι τα θεμέλια αυτής της Ένωσης ε, ισοδυναμούν με σεμβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, δημοκρατίας, κράτους δικαίου, ισότητας, ελευθερίας και σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων συμπεριλαμβανομένων και των δικαιωμάτων των μειονοτήτων. Αυτό το άρθρο πρόσφατα εισήχθη συνθήκες μόνο το 2009 και Κατά την άποψή μου αυτό σημαίνει ε, μια σημαντική μεταβατική περίοδο για την Ένωση γιατί η Ένωση παλαιότερα ήταν μια Ένωση δημοκρατιών και τώρα πλέον μεταλλάσσεται σε Ένωση Δημοκρατίας, Δημοκρατικών Αξιών. Αυτό λοιπόν το άρθρο δεν είναι ένα ε, γραφειοκρατικό πόνημα των ε, Βρυξελών ήταν μια επιλογή των κρατών μελών που επέλεξαν να συμμετέχουν όλα τα κράτη, κυρίως η Ουγγαρία. Ένα τμήμα του άρθρου 2 προτάθηκε ε, ειδικά από την κυβέρνηση αυτό δηλαδή που αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα των μειονοτήτων. Και το άρθρο αυτό εγκρίθηκε από τα κράτη-μέλη η Ουγγαρία ήταν η πρώτη χώρα που επικύρωσε τη συνθήκη της Λισαβόνας με το άρθρο 2. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι οι αξίες αυτές ε, γίνονται σεβαστές από τα κράτη-μέλη σε μια κοινωνία που είναι δημοκρατική και προσβλέπει στις ε, στο ανώτατο δυνατό επίπεδο ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ισότητα των δύο φύλων, διαφάνεια και πάρα πολλά άλλα. Νομίζω ότι αυτές είναι οι αξίες που προβάλλει και το 1999 ή στη δική μου τη χώρα το 1974. Το αίσθημα δηλαδή του να ανήκει κανείς στην Ένωση, αυτό είναι μια διασφάλιση για τους Ευρωπαίους ότι θα ε, προστατεύονται τα δικαιώματά τους και αν ε, ε, παραβιάζονται τα ανθρώπινα του ενός, παραβιάζονται τα ανθρώπινα τα δικαιώματα όλων. Η Ουγγαρία έχει να παρουσιάσει τα βάσια παραδείγματα για αυτές τις αρχές το 56, το 89. Το θέμα είναι πόσο σοβαρά λαμβάνουμε τη διατύπωση του άρθρου 2 ε, δεν υπάρχει καμία εμβολή για μας τους βουλευτές ότι τα το άρθρο αυτό πρέπει να το λάβουμε πολύ σοβαρά γιατί περικλεί τις ε, αξίες της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης και επίσης διότι κατόπιν στο άρθρο 3 βλέπουμε ότι ο πρώτος στόχος Ένωσης είναι να προάγει τις αξίες που αναφέρονται στο άρθρο 2. Δηλαδή η ευθύνη μας δεν είναι παθητική αλλά και ενεργητική ότι έχουμε το καθήκον να προάγουμε αυτές ε, τις αξίες και με βάση την αρχή της ε, συνεργασίας να άρουμε οποιοδήποτε εμπόδιο ε, σε αυτές τις αξίες, διότι οτιδήποτε άλλο υποσκάπτει την αξιοπιστία της Ένωσης. Το να λαμβάνει κανείς ε, αυτές τις αξίες ε, σοβαρά σημαίνει επίσης ότι ε, εφαρμόζουμε και μια σοβαρή μεθοδολογία. Μια μεθοδολογία που επιτρέπει διορθώσεις, προσθήκες, τροποποιήσεις και αφορά όλες τις πολιτικές ομάδες. Η έκθεση αυτή είναι μακροσκελής Βέβαια τα κομμάτια που την αποτελούν ε, είναι συνεδεμένα μεταξύ τους, γι' αυτό και καλό όλους σας ε, ή δυνατόν να διαβάσετε όλο το έγγραφο. Επιτρέψτε μου να σας πω το εξής. Στις πρώτες ε, σελίδες βλέπουμε την ερμηνεία των αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτά μοιάζουν ε, με αυτά που σας είπα και προφορικά. Βλέπετε το υπόβαθρο στην ε, έκθεση με τις ε, αλλαγές, τις νομοθετικές και συνταγματικές στην Ουγγαρία τον τελευταίο 1,5 χρόνο. Όπως γνωρίζετε έλαβαν χώρα πολλές αλλαγές, τροποποιήθηκε το Σύνταγμα, τώρα θα έχουμε ένα νέο σύνταγμα και από τη στιγμή ε, που εγκρίθηκε έχει ήδη τροποποιηθεί τέσσερις φορές. Την τελευταία φορά μάλιστα υπήρξαν εκτενείς αλλαγές. Κατόπιν έχουμε ε, νόμους ε, ε, που μπορούν να εγκριθούν μόνο με ειδική πλειοψηφία των δύο τρίτων. Αυτό μπορεί να συμβαίνει τώρα στο Ουγγρικό Κοινοβούλιο, αλλά δεν είναι σίγουρα θα συμβεί και στο μέλλον. Και υπάρχουν διάφορα σημεία, περίπου 26 νομίζω, όπου ε, το ε, Κοινοβούλιο μπορεί να ε, αποφασίσει με ειδική, όπως σας είπα, πλειοψηφία. Και υπάρχουν και άλλες αλλαγές στην ομοθεσία περίπου 500 τέτοιου είδους αλλαγές. Έχουν υπάρξει και θεσμικοί διορισμοί και άλλες εξελίξεις. Τώρα, ας κάνουμε μία αξιολόγηση. Τόσο το Σύνταγμα, όσο και οι θεμελιώδεις νόμοι αλλάζουν ουσιαστικά αυτό που αποκαλούμε ακρογωνιαίους λίθους της δημοκρατίας, δηλαδή τις προνομίες ε, της δικαιοσύνης του Συνταγματικού Δικαστηρίου. Αυτά βέβαια έχουν ε, επιπτώσεις στην κατανομή των εξουσιών. Έχουμε και μια νέα αρχή αρμόδια για τα μέσα ενημέρωσης με πολλές αρμοδιότητες. Συναντηθήκαμε με αυτή την αρχή στην ε, Βουδαπέστη. Βέβαια η αρχή αυτή τα περίπου δύο χρόνια που λειτουργεί δεν έχει παράσχει τα αντικειμενικά εκείνα στοιχεία που είναι σημαντικά για μας για να γνωρίζουμε κατά πόσον η νέα νομοθεσία έχει βελτιώσει την κατάσταση στην ε, ε, παρέμβαση, στις παρεμβάσεις ε, στη δουλειά των δημοσιογράφων, παραδείγματο χάρη. Αυτή λοιπόν η αρμόδια αρχή θα μπορούσε να δώσει κάποια, κάποιες μορφής αξιολόγηση σε ανεξάρτητους ε, παρατηρητές. Βέβαια λέμε ότι ε, χαιρετίζουμε κάποιες από τις αλλαγές που έλαβαν χώρα. Η εφαρμογή κάποιων συστάσεων δεν προχώρησε τόσο όσο πρότεινε η Επιτροπή της Βενετίας. Σε κάποιες άλλες περιπτώσεις υπάρχουν και οπισθοχωρήσεις όπως ε, το Εθνικό Δικαστικό Γραφείο Εκεί ε, συναντηθήκαμε με τον αρμόδιο δικαστή και τότε δεν ήταν σαφές κατά πόσον ο δικαστής αυτός που ορίζεται από την εκτελεστική εξουσία κατά πόσον ο δικαστής αυτός μπορεί να παραπέμπει ε, υποθέσεις ε, σε άλλα δικαστήρια κατά τη διάρκεια μιας εξέτασης μιας υπόθεσης. Εμείς βέβαια ελπίζαμε κάτι τέτοιο ε, να μην είναι δυνατόν. Είναι όμως δυνατόν, ανάλογα με τις ε, περιπτώσεις, μπορεί ο δικαστής να παραπέμπει ε, υποθέσεις ή τμήματα υποθέσεων σε άλλα δικαστήρια. Προχωρήσαμε λοιπόν σε αξιολόγηση. Χαιρετήσαμε, όπως σας είπα, τις αλλαγές. Μισό λεπτό κύριε Ταβάρης, λέει ο Πρόεδρος με κάθε σεβασμό. Έχουμε μία κοινή συνεδρίαση με την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων στις 6 παρατέταρτο. Και θα έρθουν εδώ τα μέλη της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων για αυτή την ε, συνεδρίαση για το τόσο σημαντικό θέμα την υπογραφή της Ευρωπαϊκής Σύμβασης ε, για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα έλεγα να ανακεφαλαιώσετε γιατί ε, μην ξεχνάτε ότι έχουμε και περιορισμούς, ε, χρονικούς περιορισμούς. Σας είπα, οι συνάδελφοί μας θα έρθουν εδώ σε 6 παρατέταρτο. Ευχαριστώ που μου το επισημαίνετε κύριε Πρόεδρε επειδή η δουλειά που έγινε πολύ σημαντική και κράτησε πάρα πολύ, ε, υπάρχουν και πάρα πολλέ λεπτομέρειε, αλλά εν πάση περιπτώσει θα προσπαθήσω να είμαι πιο σύντομο. Το ερώτημα που ε, έθεσα στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών την τελευταία φορά που συζητήσαμε για αυτή την έκθεση ήταν ε, διτό. Δηλαδή, πρώτον, κατά πόσον οι αλλαγές αυτές ε, είναι συστημικές ή όχι. Και στην περίπτωση που κρίνονται συστημικές, κατά πόσον πλησιάζουν τις αξίες που αναφέρονται στο άρθρο υπαριθμών 2. Η άποψη του εισηγητή είναι σαφής. Οι αλλαγές πράγματι είναι συστημικής φύσεως. Αυτό κανείς δεν το αμφισβητεί. Ε, συμφωνεί και η Ουγγρική κυβέρνηση οι αλλαγές αυτές αφορούν το δικαστικό και νομικό σύστημα στην Ουγγαρία. Όσον αφορά στη δεύτερη ερώτηση, νομίζω ότι υπάρχει γενικότερα μία τάση Βεβαίω υπήρχαν πάρα πολλές επιλογές ε, σε επίπεδο κυβέρνηση ή κοινοβουλίου. Δεν μπορούσαμε να συζητήσουμε κάθε μεμονωμένη νομοθετική διάταξη, αλλά υπάρχει έτσι ένα γενικευμένο μοντέλο ε, το οποίο απομακρύνεται αντί να ε, πλησιάζει τις αρχές που αναφέρουμε εμείς στο άρθρο υπαριθμών 2. Αυτό από μόνο του είναι ένα σημαντικό συμπέρασμα και μας βάζει σε ένα σταυροδρόμι. Δηλαδή, αν ε, λάβουμε σοβαρά υπόψη μας τις αρχές του άρθρου 2 και αν εντοπίσουμε ότι υπάρχουν συστηματικές, συστημικές μάλλον αλλαγές οι οποίες ε, οδηγούν σε απομάκρυνση από το άρθρο 2 και αν διαπιστώσουμε επίσης ότι επικρατεί μια τάση η οποία δεν θα ανατραπεί έγκαιρα, τότε πράγματι θα υπάρχει σοβαρός κίνδυνος παραβίασης ε, θεμελιωδών αξιών. Και καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι και τι έγινε, ε, δεν μπορεί να, το, να καταλήξει εκεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς ε, καταθέσαμε προτάσεις στις αρχές της Ουγγαρίας για τα θέματα που σας ανέφερα και θέλω να πω το εξής γιατί οι συστάσεις αυτές. Είναι γενικής φύσεως και δεν νομίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιθυμεί να ε, εφαρμόζονται συγκεκριμένε αρχές ε, με κάθε λεπτομέρεια. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι να γνωρίζει ότι οι αρχές αυτές είναι συμβατές με τις αρχές των συνθήκων και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι δικές μας συστάσεις κατατέθηκαν κυρίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα αναφέρω τουλάχιστον τέσσερις συστάσεις γιατί αυτές είναι και οι σημαντικότερες. Η πρώτη απευθύνεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Νομίζω λοιπόν ότι η κατακαιρματισμένη προσέγγιση που είχαμε μέχρι τώρα δεν ήταν και η πλέον κατάλληλη. Εφόσον μιλάμε για μια γενικευμένη τάση, άρα θα πρέπει να υπάρχει και γενικευμένη προσέγγιση. Εκεί που έχουμε πρόβλημα με το άρθρο 2, αυτό πρέπει να εντοπιστεί και να συζητηθεί ανάμεσα στην Επιτροπή και το κράτος μέλος. Συστήνω λοιπόν στην Επιτροπή να παρουσιάσει μια ημερήσια διάταξη με θέματα που πρέπει να εξεταστούν σε σχέση με το άρθρο 2. Δεύτερη σύσταση. Οι ευρωπαϊκοί θεσμοί δεν πρέπει να έχουν κατακαιρματισμένη προσέγγιση απέναντι στην ε, Ουγγρική κυβέρνηση. Πρέπει να συνεργαστούμε. Βεβαίως, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να έχει μια καθημερινή επαφή με την Ουγγρική κυβέρνηση αλλά και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και οι διάφορες κυβερνήσεις πρέπει να έχουν συχνή επαφή με την Ουγγρική κυβέρνηση ε, να υπάρχει ένα είδος τριμερούς διαλόγου. Αυτές είναι δύο συστάσεις συγκεκριμένες. Επειδή όμως δεν πρόκειται μόνο για την Ουγγαρία, πρόκειται επίσης για το ότι επιθυμούμε να διασφαλίσουμε να υπάρχει μια ε, συνέχεια στα κριτήρια της Κοπενχάγης, τα οποία καλούνται να σεβαστούν τα υποψήφια κράτη όταν πρόκειται να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εμείς ε, αποφασίσαμε άτυπα έστω ε, να υπάρχει καταρχήν ένας ε, μηχανισμός ε, Κοπενχάγης, ένα αποπολιτικοποιημένο όργανο που να παντρωθεί από ανεξάρτητους και αρμόδους αναγνωρισμένου βεληνικούς από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο αλλά και από άλλους οργανισμούς για να αντιμετωπιστεί αυτή η ανησυχία ε, της ε, κυβέρνησης ε, που είναι οι διπλές καταδίκες. Το Κοινοβούλιο συστήνει να συγκαλέσουμε ένα, μια συνάντηση με τα Εθνικά Κοινοβούλια, με το Ποινικό Δικαστήριο, με μη κυβερνητικού οργανισμούς για να εξεταστεί το άρθρο υπαριθμών 2, για να εξεταστεί το πώς είναι δυνατόν να υλοποιηθούν όλα αυτά που προβλέπει το άρθρο. Κύριε Ταβάρες, μιλάτε μισή ώρα τώρα και έχουμε μόνο άλλη μισή ώρα και 12 άνθρωποι θέλουν να μιλήσουν. Σας παρακαλώ, βοηθήστε μας να τελειώνουμε πριν έρθουν και οι άλλοι συνάδελφοι για την κοινή συνάντηση. Με κάθε σεβασμό είμαι σίγουρος ότι μπορείτε να τελειώνετε. 30 δευτερόλεπτα μόνο. Η δημοκρατία έχει να κάνει και με ανθρώπους που νομίζουν ότι είναι αλάθητοι αλλά δεν είναι. Και εγώ φυσικά μπορεί να κάνω λάθος και η έκθεση μπορεί να περιέχει σφάλματα. Γι' αυτό λοιπόν αγαπητοί συνάδελφοι περιμένω τη συμβολή σας για τροπολογίες και βέβαια και η Υπουργική Κυβέρνηση θέλω να σχολιάσει την έκθεσή μου διότι η δημοκρατία αυτό είναι ουσιαστικά. Πώς δηλαδή θα εξασφαλίσουμε οι διαδικασίες που έχουμε να επιτρέπουν και την λήψη διορθωτικών μέτρων. Αυτό είναι σημαντικό και στην προκειμένη περίπτωση λόγω ε, της υπόθεσης αυτής και λόγω και της έκθεσης. Θα ακούσω λοιπόν τώρα τα σχόλια των συνάδελφων και λυπούμε πολύ που μακρυγόσα τόσο πολύ. Μπράβο, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Ταβάρες. Έχουμε ένα μακροσκελή κατάλογο. 13 συνάδελφοι έχουν ζητήσει το λόγο και έχουμε μόνο μισή ώρα στη διάθεσή μας. Σας παρακαλώ, τρία λεπτά ο καθένας. Μην το ξεχάσετε. Τρία λεπτά ο καθένας θα έχετε. Να είστε λοιπόν πολύ συγκεκριμένοι. σύντομη και μέσα στο θέμα. Έγκυλ είναι ο πρώτος ομιλητής. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εξαιρετικά έχετε κατανείμει το χρόνο ότι είμαι ο τελευταίος που σήκωσε το χέρι μου και ο πρώτος που παίρνει το λόγο. Έτσι πρέπει, έτσι πρέπει να γίνεται. Λοιπόν, ήθελα να ξεκινήσω τα τρία λεπτά Ευχαριστώ τον Ρίτα Βάρες για την παρουσίαση αυτής της έκθεσης που είναι όπως είναι και που αντικατοπτρίζει και τα έγγραφα εργασίας που έχουμε συλλέξει μέχρι τώρα και αν θέλετε ε, μία εντύπωση που έχουμε αποκομίσει κάποια μέλη της Επιτροπής μας. Να πω ότι ελπίζω να έχουμε την δυνατότητα να το ξανασυζητήσουμε, να μην είναι η μόνη φορά. Πολύ συχνά έχω πει ότι αυτά τα οποία συμβαίνουν από σταγματικής και νομικής πλευράς στην Ουγγαρία κάποιοι μπορούν να τα βλέπουν ε, με τον άνθρωπο τρόπο και κάποιοι άλλοι με τον εντελώ αντίθετο. Ξεκινάμε λοιπόν ε, με κάποια επικριτική στάση αλλά από την άλλη υπάρχουν διακεκριμένοι ε, νομικοί οι οποίοι δεν πρέπει να αφισβητήσουμε αυτά που έγινονται στην Ουγγαρία όπως πολλές φορές ισχύει ε, με τα νομικά, μπορεί κανείς να τα ερμηνεύει είτε προς τη μία είτε προς την άλλη κατεύθυνση και γι' αυτό υπάρχουν δικαστήρια και ένας διάδικος κερδίζει, ένας διάδικος ιτάται. Ε, Θα αφήσω τώρα τους ε, συναδέλφους με αφορά πολιτικές ομάδες να σημάνουν τα πιο θετικά και εγώ θέλω να αναφέρω κάποιες επιφυλάξεις μου. Παραδείγματο χάρη, συστάσεις προς τις Αρχές οι οποίε φαίνονται προ μια κατεύθυνση που ουσιαστικά επιβάλλουμε στην Ουγγαρία να δώσει ε, ένα συγκεκριμένο καθεστώ, κάποιε συγκεκριμένε αρμοδιότητε στο συνταγματικό δικαστήριο. Αυτό δεν το έχουμε ξανακάνει με κάποια άλλη χώρα. Πώ θα πούμε ω Ευρωπαϊκή Ένωση σε μια χώρα πώ θα λειτουργεί το σταγματικό τη δικαστήριο, τι έρχονται θα έχει, τι ε, λειτουργεί στα επιτελεί όταν στις άλλες 26 χώρες δεν λειτουργούν τα συνταγματικά δικαστήρια κατά τον τρόπο που θέλουμε να επιβάλλουν η λειτουργία του συνταγματικού δικαστήριου της Ουγγαρίας. Αυτό, επομένως, το συγκεκριμένο, αν περάσει, δεν με ικανοποιεί. Επίσης, αυτή η αιώνια ιστορία με την αναγνώριση των εκκλησιών. 300 εκκλησίες έχουν χάσει, λέει, το καθεστώς. Εγώ δεν ξέρω να υπάρχουν 300 εκκλησίες. Όποιος ξέρει να μου πει. Σας προκαλώ. Μπορεί να υπάρχουν 300 θρησκευτικέ ομάδε που ε, αποκαλούνται εκκλησίε, αποκαλούν αυτού εκκλησία, αλλά δεν υπάρχουν 300 εκκλησίε αναγνωρισμένε. Δεν ξέρω, δεν πιστεύω ότι αυτό ισχύει και μάλλον βλέπω ότι πρέπει να σταματήσω που να είναι, ολοκληρώνω λέγοντα ότι υπάρχουν στοιχεία που δεν με ικανοποιούν, γιατί θα σήμαινε αυτό ότι ε, πηγαίνουμε σε μια κατεύθυνση που θέλουμε να επιβάλλουμε κάτι που πιστεύουμε ότι είναι δίκαιο, αλλά αν το κάνουμε, πρέπει να το κάνουμε και σε όλε τι άλλε χώρε. Αλλά αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε. Άρα το θέμα είναι να ξέρουμε τι είναι λογικό και τι δεν είναι λογικό να συμπεριλαμβάνει η έκθεση αυτή. Και λαμβάνω ότι θέλω να έχουμε τη δυνατότητα να το ξανασυζητήσουμε και φυσικά και θα καταθέσω το Βέμπερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω καταρχάς τον Ρουί Ταβάρης για τη δουλειά του. Πράγματι όλα τα έγγραφα εκπονήθηκαν ε, σε συνεργασία με όλες τις πολιτικές ομάδες θα έλεγα. Συμφωνώ με τον εισηγητή που λέει ότι πρέπει να δούμε κατά πόσον βλέπουμε συστημική προσέγγιση αλλαγές στην Ουγγαρία. Και αν αυτή η προσέγγιση αντιβαίνει τις αρχές ε, του άρθρου 2 της συνθήκης. Συμφωνώ με την εκτίμηση του εισηγητή και το γεγονός ότι αναβάλαμε την ε, σύνταξη της έκθεσης και τη σχετική συζήτηση μέχρι σήμερα, νομίζω ότι μας έδωσε και τη δυνατότητα να δούμε τις αλλαγές στο Ουγγρικό Σύνταγμα. Αυτή η περιβόητη πλέον ε, τροποποίηση εγκρίθηκε πριν από λίγους μήνες, αλλά Μιλάμε σαν να είναι μια τροπολογία αυτή η τροποποίηση, αλλά εδώ μιλάμε για μια σελίδες από αλλαγέ από τροποποίησεις. Αν η απάντηση είναι ναι, ότι είναι δηλαδή συστημική η προσέγγιση και αντιβαίνει ε, στο άρθρο 2 της ε, συνθήκης, το επόμενο ερώτημα είναι, συνεχίζουμε με όπως ε, μέχρι τώρα, business as usual, ή ακολουθούμε μια διαφορετική πλέον προσέγγιση. Ο κύριος Έγγελ λέει ότι οι ειδικέ συγκεκριμένες συστάσεις από το Κοινοβουλίο προς την κυβέρνηση δεν είναι ευπρόσδεκτες. Τι προτείνετε λοιπόν κύριε Έγγελ, τι να ζητήσουμε από την κυβέρνηση να κάνει, ώστε να δούμε τελικά ότι οι βασικές αρχές και αξίες της Ένωσης γίνονται σεβαστές. αν δεν διατυπώσουμε συστάσεις, μήπως πρέπει να κάνουμε κάτι πιο σκληρό. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Μήπως να κινήσουμε μια διαδικασία δυνάμει του άρθρου 7. Όλα αυτά πρέπει να τα συζητήσουμε μεταξύ μας. Εγώ δεν πιστεύω ότι μπορούμε να πούμε ότι όλοι κάνουν λάθος βλέπουμε ότι το Σύμβουλο της Ευρώπης, ε, η Επιτροπή της Βενετίας, οι κυβερνήσεις, όλοι αυτοί ασκούν κριτική. Άρα κάτι δεν πάει καλά και πρέπει να αντιμετωπιστεί. Και περιμένω και εγώ βέβαια να μας πείτε ποια θα είναι η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών για να προχωρήσουμε. Ευχαριστώ κύριε Βερσιά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω και εγώ, όπως προλαλήσαντες, ε, τον εισηγητή για τον τρόπο με τον οποίο έχει εργαστεί. Δεν είναι εύκολο θέμα. Και κάθε φορά που το θίγουμε στην Επιτροπή μας, ε, το νιώθουμε αυτό. Πιστεύω ότι πράγματι προσπάθησε να καταρτήσει ένα έγγραφο που μπορεί να συμπεριλάβει τις περισσότερες από τις απόψεις των σκιωδών. Δεν θέλω να στιγματίσουμε την Ουγγαρία. Αλλά πρέπει να δείξουμε ποια είναι η προσήλωση της Ένωσης στις αξίες του άρθρου 2. Είναι ένα σύμπτωμα η Ουγγαρία. Δείχνει τις εκτροπές, ε, την ολίσθηση αν θέλετε της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης ό,τι αφορά το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Γιατί, γιατί ε, είναι αν θέλετε ένα παράδειγμα η Ουγγαρία γιατί συσσωρεύει πάρα πολλά και βλέπουμε ότι για κάθε περίπτωση ε, που αφορά την Ουγγαρία μας δίνει και ένα άλλο παράδειγμα μιας άλλης χώρας ε, που δεν ε, σέβεται τη συγκεκριμένη αρχή. Επίσης πρέπει να πούμε αν η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι και αυτή προσιλωμένη στις αρχές και αξίες του εγώ από την ΚΟΕ πραγματικά ε, έχω ένα όνειρο. Το όνειρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι θεμελιώδεις ε, αξίες, οι αξίες του άρθρου 2 να προστατεύονται ή ε, να κυρώνεται η παραβίασή τους ή να είναι κατοχυρωμένες αν θέλετε όπως ακριβώς και οι οικονομικές ελευθερίες. Ευχαριστώ κύριε Μορβάκη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να μιλήσω στα Ουγγρικά εάν μου επιτρέπετε. Μήπως όλα αυτά τα έχουμε ξαναπεί, αυτό υποπτεύομαι. Η αλλαγή καθεστώτος όπως λέμε, τα είχε δει αλλιώς τα πράγματα δηλαδή. πριν τη μεταπολίτευση υπήρχαν, διδάσκονταν στα σχολεία ως αγωγή του πολίτου αφηρημένες έννοιες με σκοπό να εμποδιστεί ακριβώς οποιαδήποτε αλλαγή καθεστώτος. Αλλά υπήρχε ακόμα η έννοια του κράτους δικαίου. Έννοια η οποία ερμηνευόταν όσο ότι δεν μπορεί κανείς να κατηγορήσει τους υπεύθυνους του κομμουνιστικού καθεστώτος για κλοπές και για όλα τα άλλα όσα είχαν κάνει. Τώρα όμως βλέπουμε ότι γίνεται μια προσπάθεια κατάργηση σχεδόν ολόκληρου στις έννοιας του δικαίου. Άρα αυτές οι λεγόμενες κοινέ αξίες της Ευρώπης πρέπει να δούμε γιατί μας αρέσουν, τι, τι είναι αυτές οι αξίες και γιατί είναι η μία σπουδαιότερη από την άλλη, γιατί θα ήταν η μία σπουδαιότερη από την άλλη. Παραδείγματο χάρη η μείωση των οικονομικών διαφορών μεταξύ χωρών, η καταπολέμηση της ανέχειας, θα μπορούσαμε να γνωμοδοτήσουμε για το ρόλο των πολιεθνικών στην Ουγγαρία ας πούμε. Στην έκθεση λοιπόν εδώ, από την πρώτη παράγραφο ήδη, στο σημείο Δέλτα, στο σημείο Δέλτα λέω, λέμε ότι πρέπει να διασφαλίσουμε τη διατήρηση των αξιών της Ένωσης. Μα ερωτώ τον εισηγητή, πού γίνονται αυτές οι αξιολογήσεις ως προς το κατά πόσον γίνονται σεβαστές οι αξίες της Ένωσης. Μετά στο σημείο 4 a szerződések előtti egyenlőségét, hol van tartva Πώς γίνονται σεβαστές οι αξίες της Ένωσης λοιπόν. Υπάρχουν οι συνθήκες φυσικά και μετά υπάρχουν και οι εθνικές εφαρμοστικές ρήτρες, ε, περιφερειακές, τοπικές. Πρέπει λοιπόν να δούμε πρώτον τι λένε οι συνθήκες και έπειτα πώς μεταφέρονται εθνικά στην ε, εθνική νομοθεσία αν θέλουμε να αποφύγουμε τέτοιου είδου συμπεριφορές τι οποίε έχουν ήδη βαρεθεί και οι Ούγγρικοι που έχουν πολύ ενοχληθεί από αυτές για να υπάρξει επιτέλους μια αλλαγή. Κοιτάξτε, και εγώ είμαι σκιώδης εισηγητής και θα μιλήσω και εγώ στη μητρική μου γλώσσα για να είμαι πιο σύντομος. Καταρχήν Χαίρομαι για τη δουλειά του εισηγητή που και του εκφράζω όλη μου την εκτίμηση και το σεβασμό για το έγγραφό του, το οποίο είναι απολύτως ισορροπημένο. Δεν θέλω εδώ να επανέλθω στις κοινέ δημοκρατικές αξίες, του κράτους δικαίου και τις θεμελιώδεις αρχές και δικαιώματα. Γιατί αυτά ήδη προβλέπονται από τη βασική αρχιτεκτονική της Ένωσης και είναι όντως κοινέ συνταγματικές μας αρχές. Δεν θα τα ξαναπώ όλα από την αρχή λοιπόν, είμαστε μια δημοκρατική ένωση αλλά και μια ένωση που πρέπει να προστατεύει τη δημοκρατία. Γιατί η δημοκρατία δεν είναι απλώς ένα σύνολο, ένα συνονθήλευμα κανόνων. Όλα αυτά στοχεύουν στην προστασία αξιών, μεταξύ των οποίων και η συμμετοχή των μειονοτήτων στην νομοθετική διαδικασία. Η σύνδεση, ο συνδυασμός της μειοψηφίας με την πλειοψηφία και αυτά δημοκρατία είναι. Γιατί μια δημοκρατία δεν είναι απλώς η διακυβέρνηση από την πλειοψηφία. Ναι, φυσικά υπάρχει ο κανόνας της πλειοψηφίας, αλλά με σεβασμό και της μειοψηφίας και των ατόμων και αυτό σημαίνει ότι δικαίως προβλέπεται και από την Κοπενχάγη δημοκρατικός έλεγχος των υποψηφίων χωρών αλλά από την ένταξη και μετά δεν πάβει η προσοχή που δίνουμε στην τήρηση των δημοκρατικών διαδικασιών και αξιών. Πρέπει κάθε υποψία άνησης μεταχείρισης να διαλευκανθεί και στη συγκεκριμένη περίπτωση στην Ουγγαρία. Δεν πρέπει όμως να χρησιμοποιηθεί η Ουγγαρία σαν πρόσχημα ή μοναδικός στόχος η Ουγγαρία. Έκανε πολλές προσπάθειες για να ενταχθεί στην Ένωση και τις προσπάθειες αυτές πρέπει να τις συνεχίσει όπως και οι άλλοι εξάλλου. Δεν τελείωσε τίποτα με την ένταξη, δεν τελειώνει τίποτα με τις εντάξεις. Το είδαμε και επί τόπου όταν πήγαμε και συνομιλήσαμε με λογικούς ανθρώπους στους οποίους θέσαμε ορισμένα εύλογα ερωτήματα όπως το θέμα του πλουραλισμού, της δικαιοσύνης, το συνταγματικό δικαστήριο, το γεγονός ότι ο νόμος προβλέπει ποιος δικαστής θα σας δικάσει για ποιο παράπτωμα ή έγκλημα. Όλα αυτά είναι ανησυχητικά. Μας ξυπνούν ξεχασμένες μνήμες και τελικά ο εκλογικός νόμος ο οποίος ίσως τελικά να επηρεάσει το εκλογικό αποτέλεσμα με μη δημοκρατικό τρόπο σκέφτομαι τις επόμενες ευρωεκλογές. είχα συνεννοήσεις με την Κομισιόν και αρχίζει εδώ μια συζήτηση που θα κρατήσει πολύ καιρό. Ο κύριος Κίρκοπ, παρακαλώ. Εγώ μιλώ εκ μέρους ε, του κ. Μακεντάι για αυτήν την συγκεκριμένη έκθεση και επιθυμώ δεν θέλω να μπω στις λεπτομέρειες σήμερα, γιατί θα υπάρξουν ε, ε, ευκαιρίες να συνεχίσουμε σε αυτή την έκθεση. Αυτό όμως που θέλω να σας πω, Πρόεδρε, και σε εσά και σε άλλους στην Επιτροπή, που ε, ενδεχομένως θα έχουν κάποια πολιτική άποψη για την Ουγγαρία, είναι ότι η Επιτροπή αυτή πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτική. Προηγουμένως, όταν μιλάγαμε για τη Βουλγορία η κυρία Μάτσιερ και άλλοι μας κατέστησαν πολύ προσεκτικούς. Δεν πρέπει να μετατραπούμε σε ανακριτική επιτροπή για τα τεκτενόμενα στα κράτη-μέλη. Ούτε πρέπει να είμαστε εδώ το αποθετήριο ε, για διάφορες απόψεις σχετικά με ένα κράτος. Δεν είναι αυτή η δουλειά μας. Εάν σε ένα κράτος υπάρχουν κάποιες ε, προδιαγραφές, κάποιοι όροι που αμφισβητούνται, και σε αυτή την Επιτροπή και σε άλλες επιτροπές για το τι ας πούμε διαδραματίζεται στην Ουγγαρία ε, πάντα σε σχέση με το τι συμβαίνει σε άλλα κράτη. Αν υπάρχουν όλα αυτά τότε εγώ νομίζω πρέπει όλα αυτά τα θέματα να τα παραπέμψουμε στην Επιτροπή που σε τελική ανάλυση είναι ο θεματοφύλακας των συνθήκων και η αξιολόγηση θα γίνει από την Επιτροπή και όχι μέσα σε ένα τέτοιο πολιτικό περιβάλλον όπως αυτό που βρισκόμαστε εμείς. Βεβαίω το να γίνεται ε, αναφορά για ένα σύνταγμα αυτό δεν αρκεί. Εγώ εκπροσωπώ μια χώρα που δεν έχει καν γραπτό σύνταγμα. Τα τελευταία 30 χρόνια στην Ευρώπη ε, συνέβησαν τα τελευταία 30 χρόνια, ε, συνέβησαν ε, πολλά στην Ευρώπη και αυτά θα μπορούσαν να μας εμπνεύσουν. Υπήρξαν ανατροπές, ε, πολλές από αυτές στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη, άρα δηλαδή προφανώς στις χώρες αυτές υπάρχουν εξελίξεις, περνάνε από δεσποτικές καταστάσεις στη δημοκρατία. Και όλα αυτά πρέπει να τα κατανοήσουμε. Ε, βεβαίως ε, άλλοι ε, είμαι σίγουρος ότι έχουν πιο πολιτικές απόψεις από αυτού. Αλλά τουλάχιστον για μένα και ελπίζω ότι εκπροσωπώ και τις απόψεις κυρίας Μάκεντάρ που συμμετείχε στην αποστολή και νομίζω συνεισέφερε τα μάλα στην έκθεση. Εμείς θα εξετάσουμε πολύ προσεκτικά την έκθεση που θα συνταχθεί Σωστά αυτά απολέκτησαν, αλλά για άλλη μια φορά επαναλαμβάνω, η Επιτροπή αυτή δεν πρέπει να επιτρέψει τον εαυτό της να μετατραπεί σε ανακριτική επιτροπή. Γιατί αυτό σας είπα είναι δουλειά εκείνων που τους πληρώνουμε, δουλειά της Επιτροπής. Αυτή πρέπει να το πράξει για μας. Αυτή είναι η θέση μου, ε, κύριε Πρόεδρε. Η κυρία Μπάουα. Είμαι πολύ σύντομη. και τον υπόλοιπο χρόνο μου δώστε τον στην Κίνγκα Γκάλ. Ευχαριστώ τον εισηγητή. Πράγματι, θα αγνοούσαμε τα κριτήρια της Κοπενχάγης αν δεν ακολουθούσαμε αυτά που μας περιέγραψε για τις μειονότητες. Για την παράγραφο 60 έχω μία παρατήρηση. Μήπως θα μπορούσαμε Μήπως ε, θα πρέπει να δούμε κατά πόσον οι απόψεις Επιτροπής Βενετίας ε, υπερέχουν άλλων απόψεων. Εσείς πραγματικά πιστεύετε ότι η Ουγγαρία δεν είναι κράτος δικαίου. Το εννοείτε σοβαρά αυτό. Σας παρακαλώ να μου απαντήσετε αυτό. Και όπως είπε και ο συνάδελφος Κυρκόπ, ε, πολλές φορές ακούμε μόνο τη μία πλευρά και δεν δίνουμε καν τη δυνατότητα στην άλλη να εκφράσει και αυτή την άποψή της. After a lengthy, very unusual... Κοιτάξτε, βρισκόμαστε μπροστά σε μία μακρά και ασυνήθιστη διαδικασία σε αυτήν την Επιτροπή. Για ένα ολόκληρο χρόνο είδαμε να προβάλλονται ε, διάφορες ασυνήθιστες λύσεις, ε, πέντε έγγραφα εργασίας, η περίπτωση της Ουγγαρίας ερχόταν και επανερχόταν συνέχεια στην ημερήσια διάταξη και αυτή η έκθεση ε, πραγματικά είναι περίεργη. Έχουμε μία έκθεση πρωτοβουλίας που, είναι, που περιλαμβάνει 31 σελίδες. Εγώ σας λέω, όποτε μου επιτράπηκε να καταρτήσω έκθεση πρωτοβουλία, μου είπανε το πολύ πολύ τρει σελίδε. Περίεργο λοιπόν αυτό τώρα με τι 31 σελίδε. Και το λέω αυτό διότι είναι απαράδεκτο το να εξετάζουμε την περίπτωση της Ουγγαρίας, να εξετάζουμε διατάξεις ε, του συντάγματος, να εξετάζουμε θεσμούς και λύσεις, να τα επικρίνουμε αυτά, να ισχυριζόμαστε ότι δημιουργούν προβλήματα τη στιγμή που παρεμφερείς διατάξεις, ε, θεσμοί και λύσεις υπάρχουν και σε άλλα κρατημέλη και ποτέ δεν αμφισβητήθηκαν πόσο μάλλον να επικρίθηκαν. Εφόσον λοιπόν Αυτά που λέμε για την Ουγγαρία δεν λέγονται και για όλα τα άλλα κράτη-μέλη όπου υπάρχουν παρεμφελείς λύσεις, εγώ ε, θα ισχυριστώ ότι εδώ εφαρμόζονται δύο μέτρα και δύο διαφορετικά σταθμά. Επίσης, αυτό που είναι πρόβλημα είναι το ότι στην έκθεση αυτή επικρίνονται λύσεις οι οποίες υπάρχουν από τη δεκαετία του 90 στο ουγγρικό νομικό σύστημα. Ποτέ δεν επικρίθηκαν, ποτέ δεν αμφισβητήθηκαν και τώρα λέτε ότι οι διατάξεις αυτές είναι απαράδεκτες και ε, αναφέρομαι σε νόμους που θεσπίστηκαν με πλειοψηφία ε, δύο τρίτων. Ποτέ δεν αμφισβητήθηκαν μέχρι πρόσφατα τώρα υποτίθεται ότι όλα αυτά θέτουν σε κίνδυνο το κράτος δικαίου στην Ουγγαρία. Να πω επίσης ότι οι περισσότερες από τις 31 σελίδες παρουσιάζουν λάθη, παρουσιάζουν ισχυρισμούς και ακόμα και παραπλανητικές ερμηνείες. Και να σας πω γιατί το λέω αυτό. Γιατί αν είχε πάρει κανείς ε, σοβαρά, αν είχαν ληφθεί σοβαρά οι απαντήσεις ε, της κυβέρνησης, τότε αυτά τα θέματα που αναφέρονται στην έκθεση δεν θα αναφέρονταν, γιατί δεν ευσταθούν. Επίσης, παίρνετε τόσες, ε, τόσα πολλά αποσπάσματα από τις αποφάσεις του συνταγματικού δικαστηρίου, αλλά κατά περίεργο τρόπο ε, τα αποσπάσματα αυτά απλά αποδεικνύουν ότι υπάρχει πρόβλημα. Άλλα όμως ε, ε, αποσπάσματα ή κείμενα που δείχνουν ε, ότι ήταν απαραίτητο να ληφθούν αυτές οι αποφάσεις, αυτά δεν αναφέρονται. Άρα για μένα είναι πολύ ενδιαφέρον το πώς απομονώνει κανείς ένα κομμάτι μιας ε, απόφασης του Σταγματικού Δικαστηρίου και αφήνει όλα τα άλλα. Αυτό είναι παραπλανητικό και πολλές φορές θεωρώ ότι είναι και κακόβουλο. Και σωστά αυτό που λέτε. Δεν μπορεί εδώ η Επιτροπή να παίζει το ρόλο δικαστηρίου. Αυτό το σχέδιο έκθεσης μοιάζει να, με καταδικαστική απόφαση δικαστηρίου και είναι απαράδεκτο αυτό. Ε, διότι η άλλη πλευρά δεν έχει την ευκαιρία να εκφράσει την άποψή της, δεν έχει τη δυνατότητα να ανατρέψει ισχυρισμούς. Γι' αυτό λοιπόν... Ε, Όλα αυτά δεν είναι αλήθεια. Κατόπιν τούτου, πρόεδρε, αν ε, ήσασταν ε, γενόδρος, αν είχαμε χρόνο, θα μπορούσατε να μας δώσετε χρόνο να εξετάσουμε τα 31 άρθρα για να μας πείτε ποια άρθρα είναι άδικα και ποια όχι. Αυτό θα ήταν το σωστό. Αλλιώς δεν νομίζω ότι μπορεί να ισχυριστεί κανείς οτιδήποτε για το αξιόπιστο της συζήτησης και του ψηφίσματος. Και τώρα θα ήθελα, ναι το ξέρω αλλά αφήστε με σας παρακαλώ να ολοκληρώσω κύριε Πρόεδρε. Ας πάμε στις συστάσεις. Νομίζω ότι αυτές οι συστάσεις και ο τόνος στον οποίο είναι γραμμένες ουσιαστικά δείχνει σύγχυση ρόλων Δηλαδή ουσιαστικά υπερβαίνουμε τις αρμοδιότητες ενός κοινοβουλίου που μάλλον παραγνωρίζουμε τις ε, αρμοδιότητες ενός κοινοβουλίου και μιας κυβέρνησης που έχουν εκλεγεί ελεύθερα. Άρα αυτή η σύγχυση ρόλων είναι απολύτως απαράδεκτη. Και όλοι μας, όχι μόνο εγώ, όλοι μας ε, νιώθουμε, νομίζω σχεδόν όλοι, όσοι ακούνε τις συστάσεις αυτές, τις αντιλαμβάνονται ως ένα τελεσίγραφο προς την Ουγγαρία, που επιβάλλει πράγματα που αν τα κάνατε σε οποιαδήποτε άλλο κράτος μέλος της Ένωσης, η Ένωση θα κατέρεε αμέσως. Άρα, αυτή η μέθοδος, αυτές οι συστάσεις ε, Εάν δεν κάνετε το ίδιο και με όλα τα άλλα κράτη, μέλη, θεωρώ ότι είναι εντελώ απαράδεκτο. Πρόεδρος, παρακαλώ. Ε, να δώσω το λόγο στον κύριο Βάιντεν Φόλτσε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ είμαι από χώρα γειτονική της Ουγγαρίας, από την Αυστρία. Η Ουγγαρία είναι πράγματι η γειτονική μας χώρα που μας είναι η πιο αγαπητή. Έχουμε κοινή ιστορία και από το 56 μέχρι το 80 η ρήξη του σιδηρού παραπετάσματος κλπ. Εγώ συμπαθώ ιδιαίτερα τους Ούγγρους και πραγματικά υποφέρω από όλα αυτά που ακούμε και για το πώς εξελίχθηκε η κατάσταση. Μοιάζει να μην υπάρχει διέξοδος από αυτή τη συζήτηση η Αυστρία έζησε και αυτή στο πετσί της κυρώσεις που ήταν ε, λανθασμένες, άδικες ε, και δημιούργησαν μια κατάσταση στο εσωτερικό της χώρας μας όπου δεν μπορούσαμε να βγούμε πια από αυτό το κλουβί. Καταλαβαίνω λοιπόν ψυχολογικά το πώς εξελίσσεται η κατάσταση στην Ουγγαρία. Βεβαίως τώρα δεν είναι κατάλληλη στιγμή για να σας παρουσιάσω την πολιτική μου θέση που προφανώς και έχω και απέχει κατά πολύ από όλα αυτά που διαδραματίζονται αυτή τη στιγμή στην Ουγγαρία. Νομίζω όμως ότι η έκθεση του συναδέλφου Ταβάρες είναι σημαντική. Βεβαίω και μπορούμε να καταθέσουμε τροπολογίες, αλλά εν πάση περιπτώσει η έκθεση αυτή προσπαθεί να μην δει την κατάσταση νομικίστικα, αλλά να την αξιολογήσει. Και πραγματικά αυτό είναι μια αξιέπαινη προσπάθεια να αποφύγουμε το δίλημα, να βγούμε από το δίλημα. Γιατί υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα μεγάλο δίλημα. Εγώ λοιπόν χαιρετίζω αυτή την προσπάθεια και θεωρώ ότι αποτελεί ε, μια δυνατότητα να ξεφύγουμε από το αδιέξοδο. Ε, αυτά όλα ε, που μοιάζουν με συναγερμό, αυτά που αναφέρθηκαν, ε, θα λειτουργήσουν προληπτικά και για άλλα κράτη, ε, να ξέρουν τι μπορεί να ακολουθήσει. Και αυτό θεωρώ ότι είναι σημαντικό για μας ως Ευρωπαίους. Εξάλλου, θεωρώ ότι θα έπρεπε και το Συμβούλιο να τοποθετηθεί στο πρόβλημα. Το να μην εκφράζεται το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το βρίσκω ιδιαίτερα προβληματικό. Ευχαριστώ πολύ. Ξέρετε το πιο θλιβερό είναι ότι οι περισσότεροι Ούγγροι τα θεωρούν όλα αυτά σαν αδικία, σαν αντιουγγρική καμπάνια και πράγματι η πίστη μας στην Ευρώπη έχει τροποποιηθεί από αυτή την κατάσταση. Έχει επηρεαστεί. Δύο πράγματα λοιπόν. Κανένας δεν μπορεί να πιστέψει ότι η Ουγγαρία είναι η μόνη χώρα που αντιμετωπίζει τέτοια φαινόμενα. Ας εξετάσουμε λοιπόν όλα τα κράτη-μέλη και να δούμε αν υπάρχουν τέτοιες αναλογίες. Στην Ουγγαρία αναρωτιόμαστε πώς γίνεται την εποχή της σοσιαλιστικής κυβέρνησης εδώ και τέσσερα χρόνια, α, επί τέσσερα χρόνια να συμβαίνουν πράγματα που δεν παραβιάζουν απλώς την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία αλλά που την κατακουρελιάζουν. Θυμάμαι τον τρόπο με τον οποίο διέλυσαν διαδηλώσεις, ότι χτύπησαν παιδιά και όλα αυτά με αποδείξεις. Αλλά δεν υπάρχει κι άλλα. Πώς γίνεται δηλαδή, αν είναι κανείς τόσο ευαίσθητος στις ευρωπαϊκές αξίες, οι μυστικές υπηρεσίες να μην κάνουν τίποτα. Μιλάω μόνο για αποδεδειγμένα γεγονότα. Ο διευθυντής λοιπόν των Ουγγρικών Μυστικών Υπηρεσιών κρυφά έφερε στη χώρα Ρώσους πράκτορες για να εξετάσουν τα φρονήματα στην ουσία του πληθυσμού. Εμείς είμαστε βέβαια μέλη της Ένωσης και του ΝΑΤΟ πια και τι μπορούμε να πούμε σε εκείνους που αναρωτιούνται γιατί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν σκανδαλίζεται όταν βλέπει να χτυπούν παιδιά σε νόμιμη διαδήλωση. Υπήρξαν λοιπόν πολύ σοβαρές παραβιάσεις της νομοθεσίας και της εθνικής και της ε, ενωσιακής κατά την τετραετή αυτή σοσιαλιστική περίοδο και δεν ε, ακούστηκε τίποτα. και τώρα τα παρουσιάζουν όλα σαν απλώς καμπάνια δυσφήμισης. Και εγώ ουγγρικά θα μιλήσω κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος Σταβάρες άρχισε με την παράθεση μιας ουγγρικής φράσης. Πράγματι η πατρίδα είναι, σημαίνει δικαιώματα, αλλά κανείς δεν καταλαβαίνει τι γίνεται τελευταία. Μήπως σημαίνουν όλα αυτά ότι δεν υπάρχει πατρίς ή ότι δεν υπάρχει πια από αυτά, για αυτά που υπόθηκαν από την Επιτροπή της Βενετίας και τα λοιπά, εάν είχαμε προσέξει τα κριτήρια της Κοπενχάγης και τις συστάσεις της Επιτροπής της Βενετίας, παραδείγματος χάρη για αυτά που έκανε η Σλοβακία στη νομοθεσία της για τη γλώσσα Εγώ ήμουν μέλος της Ερευνητικής Επιτροπής για τους Ούγγρους της Ρουμανίας. Έγινε λόγος για αντισημιτισμό, γίνεται λόγος για έλλειψη ανεξιθρησκείας, αλλά δεν έγινε ποτέ λόγος, δεν βρήκαμε καμία περίπτωση τέτοιων φαινομένων στην Ουγγαρία. Διαβάστε, διαβάστε το έγγραφο, διαβάστε. Μερικοί λένε ότι υπήρξαν 300 θρησκείες. Τι, τι αριθμός είναι αυτός, εννοούν μαζί και τις μάγισσες. Υπάρχουν δημοκρατικές διαδικασίες στην Ευρώπη λοιπόν. Λοιπόν λέγω. Στην Ουγγαρία δίνονται περίπου 30 λεπτά για να μιλήσουν οι επίσημοι εκπρόσωποι του κράτους και μετά σε άλλους δίνουν μια μισή ώρα, τέλος πάντων. Ο εισηγητής ζήτησε τροπολογίες, εναμένει πάρα πολλές τροπολογίες και μάλιστα διαγραφής. Κύριε Πρόεδρε, πριν από κάποια χρόνια πήγαμε στην Ιταλία ε, για να δούμε ε, πώς ε, δακτυλοδεικτούνταν η Αθήγανοι Ρωμά από την κυβέρνηση Μπερλουσκόνη. Και ε, δυστυχώς δεν είδαμε τίποτα. Και γυρίσαμε πίσω απρακτή και η Ρωμά αποκόμισε την εντύπωση ότι απλά ήταν το μήλο της έρηδας ε, ανάμεσα σε δύο πλευρές. Εδώ γίνεται λόγος για ε, συμπεριφορές αντισημιτικές στην Ουγγαρία κατά τον Ρωμά και λέω τότε ε, στην Ιταλία δεν βρήκαμε τίποτα και τώρα στην Ουγγαρία τα αισθήματα αυτά είναι πολύ λιγότερο έντονα από ό,τι πριν από τρία-τέσσερα χρόνια. Ε, πριν από τρία-τέσσερα χρόνια μερικοί απλώς και μόνο επειδή ήταν Ρωμά τους σκότωναν, τους δολοφονούσαν. Σήμερα δεν υπάρχει πια. Βέβαια η δικαιοσύνη έχει επιληφθεί αυτών των ε, θεμάτων για να διαπιστώσει ε, μήπως είχε εμπλακεί, είχαν εμπλακεί μυστικές υπηρεσίες ε, ε, σε αυτές τις υποθέσεις. Το να ισχυρίζεται κανείς τώρα ότι βρίσκονται σε έξαρση αυτά τα αισθήματα κατά των Εβραίων και κατά των Ρωμά στην Ουγγαρία, θέλω να σας πω ότι η Ουγγαρία τα τελευταία δέκα χρόνια εργάζεται σκληρά επί του θέματος. Ε, ε, εγώ εκπροσωπώ πλέον τους Ρωμά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και δουλέψαμε σκληρά για να αποδείξουμε ότι δεν ισχύουν όλα αυτά. Εάν η Ουγγρική κυβέρνηση δεν είχε βάλει το θέμα στην ημερήσια διάταξη του 2011 του Συμβουλίου, ε, θα εξακολουθούσαμε να μην έχουμε τα εργαλεία να αντιμετωπίσουμε τον αντισημιτισμό και αισθήματα κατά τον Ρωμά. Εγώ όλα αυτά τα λέω όχι ως εισηγήτρια, αλλά όχι ως Ουγγαρέζα, αλλά και ως εισηγήτρια για ε, προγράμματα υπέρ των ε, Ρωμά, σας λέω λοιπόν ως ε, εισηγήτρια ότι το εγκουρικό δικαστήριο ή τα εγκουρικά δικαστήρια είναι τα καλύτερα. Σουηδία και Φιλανδία έπονται. Στην Ουγγαρία Πολλοί άνθρωποι περιμένουν βέβαια να αποκτήσουν τις σωστές πληροφορίες. Στην Ουγγαρία μάχονται κατά ε, αρνητικών συναισθημάτων εις βάρος των Ρωμά, των ε, Εβραίων και γι' αυτό η εκτέση είναι πολύ σημαντική. Αναφέρεται εδώ ότι το Ουγγρικό Κοινοβούλιο έχει θέσει σε ισχύ την απαραίτητη νομοθεσία δεν λέτε όμως γιατί ο Όρμπαν αναγκάστηκε να κάνει αυτό το βήμα, γιατί πριν από τον Όρμπαν υπήρχαν ε, ομάδες ε, που παρήλευαν στους δρόμους και φώναζαν ε, «Αθήγκανοι θα πεθάνετε». Τώρα πια δεν μπορεί να γίνει αυτό, απαγορεύεται. Γιατί το Σύνταγμα απαγορεύει τον, τον αποδαβλίζεται το μίσος. Ο Όρμπαν εξήγησε πάρα πολύ καλά ότι πολλές φορές η μυσαλλοδοξία προκύπτει από οικονομικά προβλήματα. Όταν οι εκθέσεις είναι προκατηλημένες, αυτό λειτουργεί εις βάρος των Εβραίων, των Ρωμά και άλλων. Και αυτό είναι ο μεγαλύτερος φόβος μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Ιντεβελτ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρέπει να πω ότι αυτή τη συζήτηση την έχουμε κάνει επανειλημμένα. Δεν οδηγεί πουθενά και συμφωνώ με εκείνους που βρίσκονται στην αριστερή αλλά και στη δεξιά πλευρά του Κοινοβουλίου ότι το θέμα δεν είναι της δικής μας Επιτροπής αλλά των αρμόδιων αρχών. Γι' αυτό λοιπόν λέω ότι πρέπει να ξεκινήσει η διαδικασία 7-1 και πρέπει να σας πω ότι απορρίπτω αιτιάσεις Ούγκρων αλλά και άλλων συναντέλφων ότι τα κίνητρά μας είναι πολιτικά, ότι υπάρχει ένα είδος ε, συνωμοσίας. Κουράστηκα πια. Ακόμα και η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών έγραψε μία επιστολή στην Ουγγρική κυβέρνηση. Μπορεί κανείς να κατηγορήσει τους Αμερικανούς για πάρα πολλά, αλλά ε, όχι ότι έχουν ε, πολιτικά κίνητρα με τον κατηγορούν τους Ούγγρους. Ούτε τον ΟΣΑ, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή την Επιτροπή της Βενετίας δεν έχουν όλοι αυτοί οι πολιτικά κίνητρα. Ε, το απορρίπτω αυτό και πρέπει πια να σταματήσουμε να μιλάμε για συνωμοσίες και να δούμε την ουσία του θέματος. Είναι σωστά τα στοιχεία στην έκθεση. Μπορεί ναι, μπορεί όχι, δεν το γνωρίζω. Έχετε όμως τη δυνατότητα να καταθέσετε τροπολογίες όπως και όλοι οι άλλοι βουλευτές. Φτάνει πια. Σταματήστε εδώ να θυματοποιήσετε. Με κουράσατε και νομίζω ότι η έκθεση Ταβάρες δίνει μια ολοκληρωμένη εικόνα. Εγώ δεν μπορώ να κρίνω τις λεπτομέρειες της έκθεσης. Και δεν νομίζω ότι μπορούμε να το κάνουμε αυτό σήμερα. Εγώ ε, θα ήθελα οι συστάσεις να προχωρούν πιο πολύ, να ξεκινήσει η διαδικασία 7-1, να φύγει το θέμα από την Επιτροπή και να σταματήσουν αυτές οι ατέρμονες συζητήσεις. Και μία τελική μου παρατήρηση. Μιλήσατε για δύο μέτρα και δύο σταθμά. Έχω πει επανειλημμένα σε αυτή την Επιτροπή, ναι, το κάναμε αυτό κατά κάποιον τρόπο, εάν θεωρήσετε ότι μέχρι τώρα δεν είχε ξεκινήσει αυτή η διαδικασία. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει να συνεχίζουμε τα λάθη του παρελθόντος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξελίσσεται. Αν δείτε το, την Ευρωζώνη, μιλάμε τώρα για πράγματα που έπρεπε να έχουμε εφαρμόσει πριν από 10 χρόνια. Αλλάζουν οι μέθοδοι στην Ευρωζώνη και πρέπει να αλλάξουν και σε σχέση με τα θεμελιώδη δικαιώματα. Γιατί είτε είμαστε ε, κοινωνία αξιών είτε όχι. Και όταν πιστεύουμε ότι υπάρχει σοβαρός κίνδυνος παραβίασης θεμελιωδών δικαιωμάτων, τότε πρέπει να δραστηριοποιούμε τα. Αν δεν έχουμε το θάρρος να το κάνουμε, να πάψουμε να μιλάμε για αξίες. Το θέμα μας δεν είναι η Ουγγαρία το θέμα είναι η δυνατότητα της Ευρώπης να υπερασπίζεται τις αξίες της. Και μια τελική παρατήρηση. Θα χαιρόμουν πάρα πολύ αν η Ευρωπαϊκή Ένωση έρχονταν στη δική μου τη χώρα, την πέρναγε μέσα από ενδελεχή έλεγχο και ναι να έβρισκε ε, περιπτώσεις γιατί η χώρα μου πράγματι παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Σας παρακαλώ, ελάτε στην Ολλανδία και σε άλλα κράτη-μέλη να πάτε και να ελέγξετε τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Κύριε Ταβάρης, θα έλεγα να είστε σύντομος γιατί έχουμε καθυστερήσει πάρα πολύ. Ναι, ναι, θα είμαι πολύ σύντομη εγώ. Πράγματι η έκθεση δεν αφορά μόνο την Ουγγαρία. Μπορεί να οδηγήσουν οι συστάσεις της στην του διλήμματος της Κοπενχάγης που συζητήσαμε πολλές φορές εδώ. Θέλω να προσθέσω όμως μερικές πληροφορίες που είναι σημαντικές χωρίς λεπτομέρειες. Δηλαδή ο νόμος για τις εκκλησίες. Δεν είναι το θέμα οι 300 ή όχι θρησκείες ή εκκλησίες. Το θέμα με τον νόμο αυτό είναι το κατά πόσον μια εκκλησία μπορεί να αναγνωριστεί ως τέτοια ή όχι και έχει πολιτικά κριτήρια μια απόφαση του Κοινοβουλίου χωρίς δυνατότητα προσφυγής. Αν το Κοινοβούλιο καθόριζε ελάχιστα κριτήρια βάσει των οποίων να μπορούν να διοδοτηθούν ή να απαγορευτούν εκκλησίες θα ήταν πιο σαφή τα θέματα. Δεν πρόκειται όμως για τον αριθμό τους. Τώρα για το αντιτσιγκανικό αίσθημα. Υπάρχει σε πολλές χώρες. Το πρόβλημα είναι ότι η Ουγγρική κυβέρνηση υποβοηθεί προσωπικότητες της ακροδεξιάς που είναι φανερά αντισημίτες και αντιτσιγκάνοι. Και το πρόβλημα πάλι είναι ο ρόλος της κυβέρνησης εδώ. Είναι λυπηρό, αλλά πάλι συνεχίζονται οι διαδηλώσεις και τα συλλαλητήρια. Μπορούμε αν θέλουμε να επισέλθουμε σε λεπτομέρειες, αλλά το όλο θέμα είναι επικίνδυνο. Υπάρχουν πάρα πολλά συγκεκριμένα προβλήματα το θέμα είναι το σύνολο τι γίνεται. Τώρα κύριε Ταβάρες τα συμπεράσματα. Α, ναι. Αγαπητοί συνάδελφοι. Κάποτε θα φύγουμε από το κοινοβούλιο όλοι. Και όταν θα επιστρέψουμε στην κανονική μας ζωή τι θα θυμηθούμε από το Κοινοβούλιο, τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις αξίες. Θέλουμε να είναι, υπάρχει ένα ενεργό Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να είμαστε σίγουροι ότι στη θέση μας θα υπάρχει κάποιος άλλος εκλεγμένος από εμά, γιατί πρόκειται για δημοκρατικά εκλεγμένο Κοινοβούλιο, που δεν θα σιωπήσει αν υπάρχουν παραβιάσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Αυτό θα ήθελα εγώ ως πολίτης από τη στιγμή που θα φύγω από εδώ μέσα. Αυτό πρέπει να σκεφτούμε όλοι όταν συζητούμε τέτοιου είδους θέματα, διότι έχουμε μια εντολή από τους πολίτες μας και θέλουμε να διασφαλίσουμε βάσει του άρθρου 3.1 ότι προωθούμε τις δημοκρατικές αξίες και για μας και για τους μελλοντικούς μας πολίτες όταν θα έχουν, έρθουν στη θέση μας άλλοι ευρωβουλευτές και θα θέλαμε και εκείνοι να φερθούν με τον τρόπο που θέλουμε να πιστεύουμε ότι πρέπει να φέρονται οι ευρωβουλευτές. Φυσικά και σε προηγούμενες θητείες υπήρχαν προβλήματα και είπαμε ότι δεν έκαναν τίποτα οι προηγούμενοι ευρωβουλευτές άρα μπορούμε και εμείς να μην κάνουμε τίποτα αλλά αυτό δεν είναι πραγματική επιλογή. Φυσικά υπάρχουν προβλήματα σε πολλές χώρες μέλη. Φοβάμαι όμως ότι αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν επιδείξει την απαραίτητη σοβαρότητα για τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τη στιγμή που μετά το 9 και μόνο υπάρχει το άρθρο που μας επιτρέπει να το θίξουμε, τότε θα πολλαπλασιαστούν αυτά. Θέλουμε λοιπόν σαν άλλα πολιτικά όργανα στην ιστορία και εμείς να φανεί ότι αποφεύγουμε τις ευθύνες μας, ότι δεχόμαστε την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε ένα τρίτο, σε ένα τέταρτο ή στη μισή ένωση. Οπουδήποτε, είτε Γερμανία, είτε Πορτογαλία, είτε στην ε, Ολλανδία, είτε στη Φιλανδία. Οι κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια έχουν το δικαίωμα να επιδεικνύουν εφευρετικότητα όπως θέλουν στην νομοθεσία τους. Μπορούν, μπορεί να αλλάξουν το καθεστώς της χώρας τους, αλλά με δημοκρατικό τρόπο προς περισσότερη δημοκρατία και διαφάνεια και πνεύμα ανοιχτό. Αν υπάρξουν δηλαδή αλλαγές των διαδικασιών να είναι προς μεγαλύτερο άνοιγμα. Γι' αυτό και εμείς στο Κοινοβούλιο αυτό θα κάνουμε για να υπάρξει περισσότερος πλουραλισμός και στη συγγραφή της έκθεσης αυτής. Σήμερα συζητούσαμε την άποψη του συγγητή. Αύριο θα γίνει άποψη της Επιτροπής και μετά του Κοινοβουλίου, μαζί με την άποψη όσων διαφώνησαν. Εάν καταφέρουμε να ταυτίσουμε ότι υπάρχει μια τάση απομάκρυνσης από τις αξίες του άρθρου 2, τότε δεν μπορούμε να παραμείνουμε σιωπηλοί. Ούτε όμως αντίθετα να δείξουμε μια χώρα με το δάχτυλο σαν μοναδικό υπεύθυνο. Γι' αυτό και εγώ έκανα δύο συστάσεις γενικότερες και δύο ειδικέ για την περίπτωση της χώρας αυτής και ζήτησα να αντιδράσει η Κομισιόν για τα γενικά έτσι ώστε να θυγεί το πρόβλημα στο σύνολο της Ένωσης. Γι' αυτό θέλησα να εξισορροπήσω τα πράγματα και αναμένω τις τροπολογίες των συναδέλφων. Τέλος, πρέπει να ευχαριστήσω τη γραμματεία και τα γραφεία τους βοηθούς των συναδέλφων που με βοήθησαν και των δικούς μου βοηθούς και όλους τους συμβούλους μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Ταβάρη, τον εισηγητή και όλα τα μέλη που συμμετείχαν στη συζήτηση και πρέπει τώρα να ανακοινώσουμε την διορία για την κατάθεση των ε, τροπολογιών. Αυτό είναι σχέδιο έκθεσης. Η ε, προθεσμία είναι 21 Μαΐου ε, μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Αυτή είναι η διορία και τώρα ε, θα έχουμε και κλεισμένων των θυρών κοινή συνεδρίαση με την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Όσοι λοιπόν ε, δεν ε, θα έχουν δικαίωμα να παρακολουθήσουν τη συζήτηση για τα επόμενα 30-35 λεπτά παρακαλούνται να φύγουν, να βγουν από την αίθουσα ήσυχα.